Με ιδιαίτερη χαρά κηρύσω την έναρξη των εργασιών της Επιτροπής μας Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αποφάσισα να αφιερώσουμε ε, το αυριανό πρωινό ε, το μεγαλύτερο τμήμα του στην ανταλλαγή απόψεων με την Επίτροπο κυρία Φερέιρα. Όπως γνωρίζετε έχουμε πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε μαζί της και αν βρούμε χρόνο στο τέλος ε, του πρωινού θα ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύντομα να μας παρουσιάσει τα βασικά συμπεράσματα της στρατηγικής έκθεσης 2019, η οποία δημοσιεύθηκε πρόσφατα που ε, συνοψίζει την εφαρμογή και την πρόοδο των προγραμμάτων 2014-2020. Η έκθεση αυτή έχει ήδη αποσταλεί ηλεκτρονικά στα μέλη της Επιτροπής μας και φαντάζομαι ότι την λάβατε όλοι σας. Επίσης, θα σας παρακαλούσα να σημειώσετε ότι θα είναι πολύ σύντομες οι αυριανές ψηφοφορίες και προτείνω η συνεδρίασή μας να αρχίσει λίγο αργότερα, δηλαδή στις 9.30. Και από τις 10 και μετά θα έχουμε την Επίτροπο για ανταλλαγή απόψεων. Μπορούμε να εγκρίνουμε το σχέδιο ημερήσιας διάταξης, όπως τροποποιήθηκε. Δεν διαφωνεί κανείς. Ωραία. Ανακοινώσεις. Έχω τη χαρά να σας ανακοινώσω, όπως έκανα και στη συνεδρίαση των συντονιστών, ότι ο μηχανισμός δίκαιης μετάβασης ε, δόθηκε επί της ουσίας ε, ε, στη δική μας Επιτροπή. Εμείς θα είμαστε καθήλια αρμόδια. Είναι πολύ στρατηγική σημασία σε αυτό το Ταμείο. Φυσικά με τη σχετική μόχλευση θα φτάσει γύρω στα 100 δισεκατομμύρια ευρώ για να φτάσουμε στην ουδετερότητα από τον άνθρακα και να απεξαρτηθούμε από τον άνθρακα. Το κείμενο αυτό θα κυριαρχήσει φυσικά στις εργασίες μας για τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Μια πρώτη συζήτηση έχει ήδη γίνει στην Ολομέλεια, στο Στρασβούργο, συμμετείχα κι εγώ και πολλά μέλη της Επιτροπής μας έλαβαν το λόγο στην Ολομέλεια και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Αύριο λοιπόν είμαι βέβαιος ότι ο μηχανισμός αυτός θα κυριαρχεί στις συζητήσεις μας με την Επίτροπο κυρία Φερέιρα. Διότι έχουμε πολλές ερωτήσεις να τις χάνουμε για τις επιλογές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά. Θυμίζω ότι στις 19 Φεβρουαρίου θα διοργανώσουμε και ένα εργαστήρι για το μηχανισμό αυτό. Ε, θέλω επίσης να σας πω ότι αύριο θα έχουμε τη διάσκεψη των περιφερειακών ε, θαλάσσιων περιοχών της ε, Ευρώπης. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ε, διάσκεψη, συνεισφέρει πάρα πολύ στους στόχους συνοχής. πρόεδρος είναι ο Ερίκο Ρώση, ε, είναι ε, ο περιφερειάρχης της Τοσκάνης και επίσης είναι και Γενική Γραμματέας και καλό όλα τα μέλη να συμμετέχουν στη συζήτηση αυτή με τις θαλάσσιες περιφέρειες. Στις 5.30 θα έχουμε και ένα κοκτέιλ γνωριμίας, όχι για να κλείσουμε τη χρονιά που έφυγε, αλλά για να ξανασμίξουμε και να είμαστε ε, ακόμα πιο αλληλέγγυοι ε, για την καινούργια χρονιά. Και να καλωσορίσουμε, να υποδεχτούμε τον καινούριο χρόνο. Εδώ στην αίθουσά μας, μετά τη συνεδρίαση. Αυτές ήταν οι ανακοινώσεις και ερχόμαστε τώρα ε, στην ημερήσια διάταξη που προβλέπει ανταλλαγή απόψεων με την κυρία Λιλιάνα Παύλοβα, αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, την οποία έχω τη χαρά να υποδέχομαι και να ξανασυναντώ. Είχαμε ήδη πάρα πολύ θετικές ε, συζητήσεις και συνεδριάσεις και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την Επιτροπή μας και για το Κοινοβούλιο γενικότερα είναι ε, εξαιρετικά σημαντική Θυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι ο θεσμός που χρηματοδοτεί μακροπρόθεσμα ε, τα έργα, παρέχει και συμβουλέ για να φτάσουμε στην υλοποίηση των στόχων μας, όπως είναι η ανάκαμψη της οικονομίας, δημιουργία θέσεων εργασία και προώθηση, προαγωγή τη συνοχής. Έχει δραστηριότητες δανειοδοτικές με δύο βασικούς στόχους, οικονομική και κοινωνική συνοχή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής παγκοσμίω. Αυτοί οι δύο στόχοι προφανώς έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την δική μας Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Για να φτάσουμε σε αυτούς τους στόχους, το άρθρο 309 της Συνθήκης προβλέπει ε, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα ε, ε, Επενδύσεων να δίνει δάνεια και εγγυήσεις για να διευκολύνει τη χρηματοδότηση έργων στις αναπτυσσόμενες περιοχές για την ανάπτυξή του. Αυτά τα θέματα λοιπόν θα μας απασχολήσουν σήμερα. Πώς δραστηριοποιείται για την οικονομική, περιφερειακή και εδαφική συνοχή η ε, ΕΤΕΠ. Πολύ πρόσφατα, τον Νοέμβρη του 2019, ο θεσμός σας ανακοίνωσε την απόφαση του να αποκλείσει από τη χρηματοδότηση οποιοδήποτε έργο συνδέεται με τα ορυκτά καύσιμα. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ως εξέλιξη. Επίσης, ε, θέσατε ένα στόχο να φτάσουμε μέχρι το 2025 στο 50% ε, των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων σας κατά της κλιματικής αλλαγής. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρία Φόντερ Λάιεν, δήλωσε ότι μέχρι το 2030 θέλει να ε, κινητοποιήσει ένα τρισεκατομμύριο ευρώ επενδύσεων έτσι ώστε να μειωθεί κατά 50% να μειωθούν μάλλον οι εκπομπέ αερίων του θερμοκηπίου. Μέχρι το 2030 όλα αυτά. Σας καλωσορίζουμε και ελπίζουμε να μάθουμε πώς αντιμετωπίζετε αυτό το νέο ρόλο σας και τις νέες προκλήσεις που έχετε. Πώς προτίθεστε να υλοποιήσετε όλα αυτά τα σχέδια για τις επενδύσεις σας έτσι ώστε να είναι εγγυημένη η αρχή της συνοχής και τα έργα αυτά να μην στρέφονται κατά κύριο λόγο προς τις πλουσιότερες περιοχές που έχουν και μεγαλύτερη δυνατότητα απορρόφησης ή προσέλκυσης επενδύσεων. Την περασμένη εβδομάδα, όπως γνωρίζετε, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρότασή της για ένα μηχανισμό δίκαιης μετάβασης. στην χρηματοοικονομική ε, αρχιτεκτονική που προτάθηκε πρωταγωνιστή η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Μετά το σχέδιο Juncker, ε, καλείστε εσείς τώρα να προσελκύσετε σημαντικές επενδύσεις για την ενεργειακή μετάβαση, η οποία επιτρέπει και στις περιφέρειες που εξαρτώνται περισσότερο από τα ορυκτά ε, καύσιμα να ε, βγουν από αυτές τις ενέργειες περιορίζοντας όσο γίνεται ε, τις κοινωνικές επιπτώσεις και τις επιπτώσεις στην απασχόληση. Έτσι ώστε όλες οι περιφέρειες στην Ευρώπη να είναι φορείς ενός νέου οικονομικού μοντέλου χωρίς άνθρακα. Όπως ανακοίνωσα και στην αρχή, ε, τη συνεδρίαση. Εμεί είμαστε αρμόδια επιτροπή επί της ουσίας για το Ταμείο αυτό της Δίκαιη Μετάβασης. Εμεί θα εξετάσουμε την νομοθετική πρόταση και η κοινή μας ε, προσπάθεια και η συνεργασία μας αρχίζει σήμερα το απόγευμα με την παρούσα συνεδρίαση. Και προφανώς θα διαρκέσει καθ' τη διάρκεια της εφαρμογής του μηχανισμού αυτού για τη δίκαιη μετάβαση. Θα ακολουθήσουν και άλλες ε, συναντήσεις όπως ήδη έχουμε συνεννοηθεί. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εσείς και το επιτολείο σας για την ανταλλαγή απόψεων ε, με την Επιτροπή μας. Ως ήθιστε ε, θα κάνετε εσείς μια εισαγωγή και στη συνέχεια οι συντονιστές θα λάβουν το λόγο και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αγαπητή Επιτροπή, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επισκέπτες αυτούς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε σε αυτή την ανταλλαγή πληροφοριών. Είναι πραγματικά η κατάλληλη στιγμή, τρέχουν πολύ σημαντικές ε, συζητήσεις και χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι κοντά σας για να εκπροσωπήσω εδώ την ΕΤΕ, που είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για τις Επενδύσεις, παρόλο που Έχω πρόσφατα αναλάβει αυτή τη θέση. Να σας πω πως είμαι αντιπρόεδρος της ε, ΕΤΕ και διορίστηκα πριν από δυόμισι μήνες μόλις. Πιστεύω όμως πως έχω ιδιαίτερη εμπειρία στα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε γιατί στην προηγούμενη μου θέση είχα εμπειρία και επίσης έχω και μεγάλη εμπειρία ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή Ρέτζι. Οπότε ελπίζω πως θα καταφέρω να συνεισφέρω στη σημαντική αυτή συζήτηση που θα γίνει σήμερα. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με μια σύντομη εισαγωγή με κάποια βασικά δεδομένα και στοιχεία για όσους δεν γνωρίζουν ε, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, παρόλο που οι περισσότεροι σίγουρα είστε εξοικειωμένοι με το έργο της, ε, αφήστε μου αυτή λοιπόν την ευκαιρία για να μοιραστώ μαζί σας κάποια από τα βασικά δεδομένα που σχετίζονται με την τράπεζα αυτή. Γιατί ίσως δεν γνωρίζετε όλοι πως η ΕΤΕ και ο όμιλος ΕΤΕ δεν αποτελείται μόνο από την τράπεζα, αλλά επίσης από το Ταμείο Ευρωπαϊκών Επενδύσεων και ο ο όμιλός μας είναι ο μεγαλύτερος ε, δανειστής ε, πολυμερής, ε, αλλά και πιστωτής παγκοσμίω. πιο πολύ και από την Παγκόσμια Τράπεζα. Την τελευταία δεκαετία αυτή έχουμε αναλάβει έργα για πάνω από 60 δις ευρώ. Και μπορώ να σας πω ότι πολλές φορές έχουμε ξεπεράσει και τα 60 δις ετησίως. 1,2-3 εκατομμύρια ευρώ έχουμε επενδύσει τα τελευταία 60 χρόνια στις 12.000 λοιπόν έργα σε 60 χώρες και επειδή χρηματοδοτούμε περίπου το 1 τρίτο κάθε έργο κατά παράδοση, εμείς έχουμε μοχλεύσει επενδύσεις ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ από τη στιγμή που συσταθήκαμε το 1958. Είμαστε μοναδικοί γιατί όλη η πραγματογνωμοσύνη που χρησιμοποιούμε βρίσκεται υπό την ίδια στέγη, το, το οποίο σημαίνει ότι δεν χρειάζεται εξωτερική ανάθεση. Έχουμε οικονομολόγους, μηχανικούς, ε, περιβαντολόγους και η πραγματογνωμοσύνη αυτή είναι απαραίτητη όταν αντιμετωπίζουμε τις βασικότερες προκλήσεις της σύγχρονης εποχής και κυρίως εδώ μιλάμε για τη μείωση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, τη μείωση της εσωτερικής συνοχής και της εδαφικής συνοχής, αλλά και της κοινωνικής συνοχής συνάμα. Και βέβαια κυρίως η πρόκληση του περιβάλλοντος που αυτή τη στιγμή αποτελεί ένα από τα κορυφαία ζητήματα ε, του θεματολογίου μας. Ε, στη χρηματοδότηση για το κλίμα είμαστε στην κορυφή του κόσμου και το 2016 έχουμε επενδύσει περίπου 71 δις δολάρια. Και λέω δολάρια γιατί με τον τρόπο αυτό υπολογίζεται μετά τη συμφωνία για τη δράση για το κλίμα ε, ε, στο Παρίσι και έχουμε και τα πράσινα ομόλογα τα οποία εκδίδουμε για να προωθήσουμε τέτοιου είδους επενδύσεις μέχρι στιγμής και από το 2007 που τα ξεκινήσαμε έχουμε χορηγήσει ε, τέτοια ε, πράσινα ομόλογα ύψους 26 δις από το 2007. Παράλληλα, ε, χρηματοδοτούμε και τη συνοχή. 30% του δανεισμού πάει κυρίως σε έργα συνοχής. Προσωπικά για μένα, επειδή είμαι αντιπρόεδρος επικεφαλής ε, του θέματος αυτό και επιτηρώ την ε, πολιτική για τη συνοχή, για τις μεταφορές και τη συμβουλευτική, είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τη συνοχή και πως το ποσοστό αυτό θα συνεχίσει να ισχύει και για το μέλλον έτσι ώστε να είναι επαρκής η χρηματοδότηση για την πολιτική συνοχή. Χρόνο με το χρόνο λοιπόν συνεχίζουμε και εστιάζουμε τα δάνειά μας προς όφελος της ε, πολιτικής συνοχής γνωρίζοντας ποιες είναι οι ανάγκες του κλάδου και βέβαια πρέπει να σας πω πως το κλίμα είναι ε, ένας από τους χώρους στους οποίους αφιερώνουμε ιδιαίτερη χρηματοδότηση. Περιφερειακή πολιτική, πολιτική συνοχής, ποια είναι η προσέγγισή μας. Να σας πω καταρχήν πως ορίζεται αυτή από τρεις εκτιμήσεις. Όγκος, ποιότητα και επιπτώσεις. Όταν μιλάμε για όγκο, σας είπα πως είναι το 30% όλων των νέων ε, επιχειρήσεών μας, ε, συνοχή λοιπόν με περιφερειακή διάσταση και σε αιτήσια βάση έχουμε πετύχει το στόχο αυτό και πρέπει να σας πω πως πραγματικά ε, έχει τοποθετηθεί στη βάση των δράσεων μας. Από το 18, συγγνώμη, από το 2008 μέχρι το 2018 ο δανεισμός για τη συνοχή έφτασε τα 240 ε, δις ευρώ που είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Έχουμε χρηματοδόσει ε, και πολλά ε, έργα που αποτελούν κομμάτι της συγχρηματοδότησης της πολιτικής αυτής, έτσι ώστε να χρησιμοποιούμε τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για να καλύπτουμε τις υποχρεώσεις χρηματοδότησης κρατών μελών. Και από το 2007 και μετά έχουμε δώσει 30 δις περίπου δάνεια στις χώρες, στα, στις ανατολικές και νότιες περιοχές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τους στόχους μας από το 2020 και μετά θα ε, χρηματοδοτούμε ε, ε, project ανάλογα με τις νέες αποφάσεις που θα παρθούν στα πλαίσια των νέων στόχων της, των μακροπρόθεσμων δημοσιονομικών προοπτικών. Οπότε εμείς θα στηρίζουμε εθνική, χρηματοδότηση, εθνική συγχρηματοδότηση στις περιοχές συνοχής εφόσον αυτό σε πολιτικό επίπεδο αποφασιστεί. Και θα το κάνουμε σε όλους τους κλάδους όπου υπάρχει ανάγκη. Αφήνοντας λοιπόν το πρώτο και περνώντας το δεύτερο που είναι η ποιότητα, εάν χρειάζεται σημειοποιήσει την ΕΤΕ, ο πελάτης θα λάβει όλο το πακέτο. Όχι μόνο την ελάχιστη χρηματοδότηση για να καλύψει την συγχρηματοδότηση ή την ε, ε, έναρξη του έργου, αλλά και τη δική μας συμβουλευτική. Γιατί έχουμε μηχανικούς, όπως σας είπα, οικονομολόγους που αξιολογούν κάθε έργο το οποίο χρηματοδοτείται από εμά. Οπότε αν δανειστείτε από εμά, θα λάβετε επίσης και την βεβαιότητα πως ε, είναι τεχνικά και τραπεζικά βιώσιμο και στέρεο το έργο, δεν κάνουμε εξωτερική ανάθεση της αξιολόγησης και της διαδικασίας. Η αξιολόγηση γίνεται στο εσωτερικό της τράπεζας. Και από όλες τις πλευρές. Κάθε ένα, αν κρυθεί απαραίτητο, συμπληρώνεται με την συμβουλευτική που παρέχουμε. Έχουμε ένα, μια ισχυρή ομάδα συμβούλων στην τράπεζά μας, που προσφέρει την πλήρη κλίμακα πραγματογνωμοσύνης που μπορεί να χρειαστεί από κάποια χώρα. Πολύ σημαντικό αυτό για τις χώρες συνοχής, όπου το δυναμικό για να εφαρμοστούν αυτά τα έργα δεν είναι αρκετά εξελιγμένο. Τρίτον, επιπτώσεις και ε, πρόσθετη αξία παρακολουθούμε το κατά πόσο δρά καταλητικά η χρηματοδότησή μας, το κατά πόσο μοχλεύονται νέα κεφάλαια, δημιουργούνται θέσει εργασία και προωθείται γενικότερα η οικονομική ανάπτυξη. Στις χώρες συνοχέ, οι υποεπενδύσεις είναι ακόμα πρόβλημα. Ο κοινός μα στόχος λοιπόν είναι να βρούμε ακριβώς τα χρήματα για τις προτεραιότητες στο δανεισμό, να δοθούν οι εγγυήσεις και να λάβει τα χρήματα αυτά και να κινηθεί η πραγματική οικονομία. Αυτή θα είναι η βασική μας στόχη και ίσως θα πρέπει να κλείσω λέγοντας πως η ΕΤΕ πραγματικά είναι μεγάλος και καλός παίκτη στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση γιατί ε, το δικό μας χρήμα δουλεύει και δεν είναι χρήματα των φορολογουμένων, είναι χρήματα που εμείς βρίσκουμε από τους επενδυτές μας και στις αγορές κεφαλαίων. Είμαστε πάρα πολύ αποτελεσματική. Χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά τις ευρωπαϊκές, ε, τα ευρωπαϊκά κονδύλια στα πλαίσια των ευρωπαϊκών πολιτικών, των πολιτικών που εσείς εδώ διαμορφώνετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εμείς ακολουθούμε. Εμείς δεν διαμορφώνουμε πολιτική, εμείς ε, δεχόμαστε κατευθύνσει και τις ακολουθούμε. Τώρα για την Πράσινη Τράπεζα που είναι η Τράπεζα για το Περιβάλλον, θα ήθελα να πω και εδώ δύο λόγια. Είπατε κι εσείς κύριε Πρόεδρε στην εισαγωγή που κάνατε, πρόσφατα ξεκινήσαμε μια μετάβαση, μια μεταλλαγή έτσι ώστε να γίνουμε μια πράσινη Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Και τον περασμένο μήνα πραγματικά ε, ακολουθήσαμε ε, όλες τις προκλήσεις που παρουσιάζει για μας το κλίμα. Η πράσινη Ευρώπη, ε, το ε, πράσινο σύμφωνο, το Green Deal που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, είναι το πιο φιλόδοξο σχέδιο που έχει παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εμείς ως κομμάτι των δεσμεύσεων που έχουμε αναλάβει αυτή τη στιγμή θα καθελκύσουμε το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα που έχουμε χρηματοδότηση αυτών των έργων. Είμαστε το μοναδικό τέτοιο ε, χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και οι στόχοι μας είναι ξεκάθαροι. Θέλουμε να αυξήσουμε το μερίδιο ε, της χρηματοδότησης που πάει σε project υπέρ του περιβάλλοντος που είναι ε, οικολογικά βιώσιμη να είναι το 50% των δράσεών μας μέχρι το 2025 ένα 3 ευρώ θέλουμε να στεγανοποιήσουμε παγκοσμίω για τις επενδύσεις αυτές μέχρι το 2030 θα χρηματοδοτήσουμε την μετάβαση σε μία μετά τον άνθρακα εποχή στην ευρωπαϊκή βιομηχανία. Θέλουμε την οικονομική αναγέννηση έτσι ώστε πολλά από αυτά τα project να γίνουν ε, υποστηρίξιμα και βιώσιμα σε τραπεζικό επίπεδο. Και επίσης για το μηχανισμό της δίκαιας μετάβασης θα κάνουμε ό,τι μας αντιστοιχεί όπως ακριβώς ανακοίνωσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποιος είναι ο στόχος μας. Είναι ένας στόχος ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί εμείς θα εξακολουθούμε μέσω του Invest EU να έχουμε πρόσβαση στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Επίσης την εντολή για τον εξωτερικό δανεισμό, αυτή τη χρειαζόμαστε και είναι σημαντική για μας, γιατί είναι ένας τρόπος για να παραδώσουμε περισσότερα και καλύτερα και για να συγχρηματοδοτούμε τα εργαλεία και τις επενδύσεις ε, μέσω των Ευρωπαϊκών Διορθωτικών Ταμείων. Όλα αυτά είναι φυσιολογικά, γιατί η προτινόμενη δική μας στόχη και η προτεραιότητα του ευρωπαϊκού ε, προϋπολογισμού είναι απολύτως ε, συμβατή και βέβαια το ε, τελικό συμβιβασμό για τις πολιετής δημοσιονομικές προοπτικές θα πρέπει να λάβει υπόψη και τα εντός και τα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ως δεσμεύσεις του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού τμήμα των 100 δις που είναι κομμάτι του πακέτου της δίκαιης μετάβασης και του σχετικού μηχανισμού ή ΕΤΕ και το υπόλοιπο όμιλος μέσω του Ταμείου ε, Επενδύσεων θα μοχλεύσει μεταξύ του 21 και του 27 30 δις ευρώ. Έχουμε πολλά χρόνια εμπειρίας ε, έχουμε στηρίξει τη μετάβαση, την αναδιάθρωση σε περιοχές με εντατική χρήση άνθρακα, με, έργα υπέρ του περιβάλλοντος και επίσης με τον εξυγχρονισμό και την αστική ανάπτυξη. Ε, είναι κάτι το οποίο θα συνεχίσουμε υπό το μηχανισμό αυτό της δίκαιης μετάβασης και πιστεύουμε πως έχουμε το δυναμικό για να στηρίξουμε και με τις επενδύσεις αυτές να συνεχίσουμε βασιζόμενοι στην τρέχουσα εμπειρία. Αν θέλετε μπορώ να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Να σας πω τι είδους έργα αυτή τη στιγμή έχουμε εφαρμόσει. Για παράδειγμα, με το Δήμο του Κατόβιτσε. Τα τελευταία χρόνια συνεργαζόμαστε Έχουμε δανείσει πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ έτσι ώστε να έχουμε μια επιτυχή μετάβαση από πόλη ανθρακορίχων σε ένα όλο ζωντανια αστικό κέντρο, το Κατόβιτσε, το οποίο προσφέρει πολλές επιχειρηματικές ευκαιρίες πια και όπου το περιβάλλον είναι πολύ πιο υγιές για τους πολίτες. Από την Πολωνία, άλλο ένα παράδειγμα, στο Βόλμπριχ χρηματοδοτήσαμε την αναγέννηση ε, του αστικού ιστού με ε, μέτρα εξοικονόμησης ε, ενέργειας. Έχασε ένα κομμάτι του πληθυσμού τους η πόλη αυτή όταν έκλεισαν τα ορυχεία και εκεί επενδύσαμε πολύ στη στήριξη την αναγέννηση της ίδιας της πόλης. Στο Βραδεμβούργο επίσης επενδύσαμε πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ ε, για ε, τα ανθρακοριχεία, τη μετατροπή αυτών, για επιχειρήσεις ε, και για να ξεφύγουμε από το παράδειγμα των παραγωγών λιγνίτη, να σας πω τι κάναμε στο Βουκουρέστι που έχουμε 60 δις ε, ευρώ για την εξοικονόμηση ενέργειας από ε, κτίρια με ε, στόχο την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργεια από όσους ζουν στην πόλη αυτή. Και τέλος, να σας υπενθυμίσω πως προσφέρουμε και συμβουλευτικές υπηρεσίες, Τζάσπερ, Σίσπερ Ελένα, όλα αυτά τα προγράμματα έχουν ένα κομβικό ρόλο που έχουν παίξει στη διαμόρφωση της στρατηγικής μετάβασης και στα σχετικά σχέδια που έχουν ε, ε, μοχλεύσει ιδιωτικές επενδύσεις. Να σας πω για τον Τζάσπερ ότι ως εργαλείο έχουμε στηρίξει ε, πρωτοβουλίες στις περιοχές που είχαν λιγνητομονάδες και βοηθήσαμε με συμβουλευτική να εντοπίσουμε έργα, να τα ε, μελετήσουμε, να τα εφαρμόσουμε και όλα αυτά είναι σημαντικά. Ειδικά τώρα που τα κράτη-μέλη θα χρειαστούν να αναλάβουν ένα πολύ ιδιαίτερο και σημαντικό ε, έργο που είναι η προετοιμασία των εθνικών στρατηγικών μετάβασης όπου θα χρειαστεί να εντοπίσουν καταρχήν ποια θα είναι αυτή η στρατηγική και κατά δεύτερον να προετοιμάσουν τα ε, τραπεζικά βιώσιμα και όριμα έργα, τα οποία μετά θα πρέπει να τρέξουν. Εκεί λοιπόν θα έχουμε, θα έχουμε τεχνική βοήθεια, συμβουλευτική, πραγματογνωμοσύνη και για την προετοιμασία αφενός στρατηγικής και για την προετοιμασία των ίδιων των έργων αφετέρου. Και για μένα αυτό είναι ένα σημαντικό εργαλείο το οποίο προσφέρει και δίνεται να προσφέρει η τράπεζα σε μια κομβική στιγμή για όλα τα κράτη-μέλη, για τις περιοχές ε, σε μετάβαση, γιατί βρισκόμαστε σε μια στιγμή αποφασιστική. Πώς θέλουμε εμείς να επιτύχουμε αυτούς τους τόσο φιλόδοξους στόχους. Γιατί αν ο σχεδιασμός είναι σωστός, ε, μόνο τότε θα καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει. Και για να το και για να κλείσω το θέμα, εμείς στην τράπεζα ε, έχουμε μια παράδοση. Παραδίδουμε αυτά αποτελέσματα σε καινοτόμες και καινούριες ε, ε, στρατηγικές, όπως το ΕΦΣΙ για παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Αυτό Ταμείο για τις Επενδύσεις το λεγόμενο σχέδιο Juncker, το οποίο ε, παρουσιάσαμε το 2015 έτσι ώστε να έχουμε επενδύσει στην Ευρώπη και σήμερα βλέπουμε πόσο εντυπωσιακό ήταν ο αντίκτυπος των όσων κάναμε. Ίσως δεν τα προωθούμε αρκετά, αλλά σήμερα θα πω δύο λόγια. «460 δις επιπλέον επενδύσεις στην Ευρώπη έχουμε μοχλεύσει μέχρι σήμερα» και μέχρι το 22 οι επενδύσεις μας θα αυξήσουν το ΑΕΠ κατά 1,8% και θα προσθέσουν 1,7 εκατομμύριο θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Πάνω από ένα εκατομμύριο μικρομεσαίες επιχειρήσεις ήδη ωφελούνται από την αυξημένη πρόσβαση ε, σε ε, κεφάλαια μέσω των επενδύσεων αυτών, οπότε βασιζόμενοι στην εμπειρία που έχουμε αποκτήσει, βασιζόμενοι στα διδάγματα που λάβαμε από αυτή την πρωτοβουλία, πιστεύουμε πως θα αναβαθμίσουμε τις επιδόσεις μας βασιζόμενοι στην εμπειρία μας, όχι μόνο για τις νέες προτεραιότητες που τώρα προτείνονται προς ε, χρηματοδότηση υπό το InvestEU, αλλά και στις προτεραιότητες στα πλαίσια του Green Deal και οριζόντια. Οπότε ναι, θα χρησιμοποιήσουμε το όσα έχουμε μάθει μέχρι σήμερα. Μια φορά ακόμα να σας ε, διαβεβαιώσω πως η τράπεζα είναι πραγματικά αφοσιωμένη στο ρόλο αυτό, τον τόσο δραστήριο, τον οποίο έχουμε αναλάβει με πολύ ενεργό τρόπο, δίκαια μετάβαση και όπως είπατε και εσείς, εσείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά σας περασμένη εβδομάδας για το Ευρωπαϊκό ε, Πράσινο Σύμφωνο ε, είπατε διάφορα και εμείς θα σας ε, συνδράμουμε, θα σας στηρίξουμε, θα χρηματοδοτήσουμε και θα βοηθήσουμε και τα κράτη-μέλη να σχεδιάσουν και να συντάξουν αυτά τα σχέδια βασιζόμενοι στην εμπειρία μας και πάντα σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, συζητώντας πάντα την κατηγοριοποίηση και τις προτεραιότητες ε, αυτών των πολιτικών. Για την ε, πολιτική συνοχής και για την περιφερειακή πολιτική, εκεί θα επιδιώξουμε να εξασφαλίσουμε πως όλες οι επενδύσεις που θα είναι για πράσινα έργα, που θα είναι για το περιβάλλον, να χρησιμοποιήσουν τις καλύτερες συνέργειες με συμπληρωματικότητα μεταξύ χρηματοδότηση για το κλίμα και χρηματοδότηση για την περιφερειακή και συνοχ... Ε, πολιτική και πολιτική συνοχή. Σε βασικέ ε, υποδομέ, για παράδειγμα, που σε πολλέ περιπτώσει σε περιοχέ συνοχή ακόμα είναι απαραίτητε. Θα σταματήσω εδώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Συζήτηση τώρα, Νοβακόφ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Παυλώα για αυτήν την εξαιρετική παρουσίαση και ευχαριστώ πολύ και όλους τους συναδέρφους του ΕΛΚ που είναι εδώ. Τόσο πολύ άριθμοι και σίγουρα θα συμμετάσχουν στη συζήτηση και αυτή. Εγώ θυμάμαι στην προηγούμενη Ολομέλεια στο Στρασβούργο όπου η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία βρισκόταν παντού στον αέρα, στα πάντα. Η Πράσινη Συμφωνία ήταν κάτι που συζητιόταν παντού. Και εγώ στηρίζω την Πράσινη Συμφωνία, όλες τις πολιτικές που προστατεύουν το περιβάλλον και που προσφέρουν ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης για τα παιδιά, για τους νέους, τους μεγαλύτερους. Όμως ξέρω ότι τέτοιες μεγάλες μεταρρυθμίσεις απαιτούν μερικές φορές χρόνο, προσπάθεια, μεγάλη προσπάθεια και πρέπει με το μαλακό να τις χειριζόμαστε. Δεν χρειαζόμαστε επαναστάσεις όταν πρόκειται για το κλίμα, αλλά μια σταθερή εξέλιξη σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές που επέδυσαν πολλές προσπάθειες για να αναπτύξουν τις κοινωνίες μας. Ναι, μερικές φορές και έχοντας άνθρακα, ναι, πράγματι. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θέλει να αλλάξει τα πράγματα. Και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο του έργου τους, εγώ αναρωτιέμαι, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πώς θα βρει την ισορροπία να στηρίξει τις αναπτυξιακές πολιτικές της Ευρώπης αλλά και την Πράσινη Συμφωνία. Γιατί πιστεύω ότι μπορούν να συνεπάρξουν και τα δύο. Και δεν χρειάζεται να εγκαταλείψουμε το ένα τις υποδομές, για παράδειγμα, ή τη γεωργία. Δεν είναι κάτι που είναι από τη μια μεριά, όπως επίσης το αέρασμος και τα λοιπά και από την άλλη πράσινη συμφωνία. Εσείς λοιπόν πώς θα πετύχετε τη συμφωνία ανάμεσα σε αυτά τα δύο, αυτές τις δύο προτεραιότητες. Ευχαριστούμε. Για να είναι πιο ζωντανή η συζήτηση, ε, παρακαλώ απαντήστε τώρα στον κύριο Νόβακοφ ώστε να υπάρχει έτσι μια πραγματική ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα σε εσά και τους ευρωβουλευτές. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ κύριε Νοβακόφ. Ναι, πράγματι η Πράσινη Συμφωνία και η στόχοι μας, ναι, είναι πράγματα τα οποία φυσικά όλοι στηρίζουμε. Από την άλλη, ναι, δεν χρειαζόμαστε επανάσταση, χρειαζόμαστε μια εξέλιξη. Χρειαζόμαστε μια σαφή στρατηγική για το πώς θα πετύχουμε τους στόχους μας με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην ξεχάσουμε κανέναν στην πορεία. Αυτό είναι που λέω εγώ συνέχεια και είναι το μήνυμά μου που θέλω σε αυτό να επιμείνω ξανά και ξανά. Οπότε, η ενεργειακή μετάβαση ε, σίγουρα θα κοστίσει, συγχρόνως θα αποτελέσει και μια μεγάλη ευκαιρία για όλους εμάς στην Ευρώπη. Οπότε δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο το τίμημα που θα πληρώσουμε, πρέπει να το βλέπουμε και σαν μια ευκαιρία για να επανασχεδιάσουμε τα ενεργειακά μας μοντέλα. Είναι πιστεύω εγώ μια ιστορική σημασία ευκαιρία. Δεύτερον, χρειαζόμαστε χρόνο και χρειάζεται να οργανωθούμε με τέτοιο τρόπο ώστε η μετάβαση να γίνει ήπια. Όλες οι περιφέρειες, όλος ο κόσμος να νιώθουν ασφαλείς, να είναι προετοιμασμένοι, να έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα και να μπορούν να στηρίξουν τη μετάβαση αυτή στις περιφέρειες. Όπως ε, ήδη είπα και στις αγωγικές μου παρατηρήσεις, οι φιλοδοξίε μας στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι να αντιμετωπίσουμε και να ενισχύσουμε τις επενδύσεις μας ώστε να φτάσουμε στο 50% για το κλίμα και το περιβάλλον. Συγχρόνως όμως θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την συνοχή, την σύγκληση των περιφερειών με 30%. Αυτό σημαίνει ότι θα προσπαθήσουμε όσο γίνεται περισσότερο να υπάρχει μια συμπληρωματικότητα ανάμεσα στη φιλοδοξία μας για την ενέργεια και το κλίμα και από την άλλη μεριά για τη συνοχή που είναι αναγκαία για τις χώρες συνοχής και για τις ε, περιφέρειες σε μετάβαση. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή να δούμε σε κάθε έργο Ποιο είναι το πράσινο στοιχείο. Σε άλλο έργο μπορεί να είναι 2%, αλλού μπορεί να είναι 50%. Αλλά τελικά θα πρέπει να προσπαθήσουμε και θα ελέγξουμε ώστε να υπάρχει σωστή ισορροπία ώστε στο τέλος της 7ης χρονιάς να έχουμε πετύχει αυτή την ισορροπία, να έχουμε δηλαδή όλο και περισσότερο την πράσινη διάσταση σε κάθε πρόγραμμα συνοχής. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα έχουμε 50% σε όλα. Σε άλλο θα έχουμε 2, σε άλλο θα έχουμε 60%. Δεν ξέρω, θα δούμε ανάλογα με τις ανάγκες. Γι' αυτό είπα ότι είναι πολύ σημαντικό για κάθε χώρα όταν αναπτύσσουν τις εθνικές τους στρατηγικές να λάβουν υπόψη τους αυτή την μετάβαση και ετοιμάζοντας τα επόμενα προγράμματά τους να σκεφτούν πώς και με ποιο τρόπο θα τα σχεδιάσουν και πώς θα στηρίξουν τις περιφέρειες σε μετάβαση, κοινωνική και οικονομική από τη μια και από την άλλη πώς θα στηρίξουν την ενεργειακή τους μετάβαση. Εμείς είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε και την ενεργειακή μετάβαση, αλλά και την ε, οικονομική ανάπτυξη των περιφερειών, της μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις διάφορες βιομηχανίες, ώστε τους διάφορους κλάδους, ώστε να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όπως είπα, δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε κανέναν, ούτε περιφέρεια, ούτε και ανθρώπους. Κυρίως αυτοί που ζουν εκεί που υπήρχαν ανθρικορυχεία. Δεν πρέπει να τους ξεχάσουμε. Πρέπει να είναι σε θέση οι άνθρωποι αυτοί να παραμείνουν στη γη τους. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία και σίγουρα είναι μια πρόκληση. Πάντως προς το παρόν εμείς στην τράπεζα είμαστε σε μια διαδικασία προετοιμασίας της αναθεώρησής μας για τους κανόνες επιλεξιμότητας και για το πώς θα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά που προτείνονται προς υιοθέτηση. Φιλοδοξία μας είναι να πετύχουμε την ισορροπία, τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην πολιτική συνοχής αφενός και την δικαιωτή μετάβαση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ε, για τους σοσιαλιστές, Μάρκες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Παύλοβα, ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Θα ήθελα να ξεκινήσω αναφερόμενος στη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την χρηματοδότηση της νέας αυτής προτεραιότητας που έχουμε στην Ευρώπη. Η τράπεζα προσπαθεί όλο και περισσότερο να γίνει μια κλιματική τράπεζα. Κάτι το οποίο βέβαια πηγαίνει χέρι-χέρι με την προτεραιότητα συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σωστό αυτό. Θα ήθελα συγχρόνω να πω ότι πιστεύω ότι η τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έχει να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην πιο κρίσιμη στιγμή τη κρίση. Να στηρίξει τι δημόσιε επενδύσει και όπω είπατε κι εσεί, σε πολλέ περιπτώσει το εθνικό κομμάτι επενδύσεων με ευρωπαϊκά κονδύλια. Είναι πολύ καλό που είχαμε την χρηματοδότηση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων του Εθνικού Κομματιού. Τώρα ξέρουμε, το περιβάλλον έχει αλλάξει. Η αγορά έχει αλλάξει και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σήμερα λειτουργεί μέσα σε μια κατάσταση όπου υπάρχουν περισσότερα χρήματα διαθέσιμα στην αγορά, πιο φτηνά ακόμα και για τις χώρες μέλη, για τις εθνικές κυβερνήσεις. Συνεπώς, ο κανόνας που μπορεί να εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σήμερα μπορεί να διαφοροποιηθεί από εκείνον που είχε τη χειρότερη στιγμή της κρίσης. Χρειαζόμαστε περισσότερο από ένα τρεις επενδύσεις για να διασφαλίσουμε την μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία και μια πράσινη κοινωνία. Εμείς συμφωνούμε με το 1-3, αλλά πιστεύουμε ότι χρειάζονται συνολικά πολύ περισσότερα αν θέλουμε να πετύχει αυτή η μετάβαση, να είμαστε και ανταγωνιστικοί αλλά και δίκαιοι. Και όπως είπατε, το θέμα της μετάβασης στις περιφέρειες που θα επηρεαστούν περισσότερο, στις περιφέρειες που ήδη είναι συνοχής, καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση εκεί είναι κρίσιμη. Και για να είμαι ειλικρινή, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πιο δημιουργικοί, να βάλουμε τη φαντασία μας να δουλέψει περισσότερο για να πετύχουμε τους στόχους χρηματοδότησης της οικονομίας και των περιφερειών αυτών. Εγώ Ήμουν υπεύθυνο ω υπουργό για την χρηματοδότηση τη χώρα μου και ξέρω ότι είχαμε πάρα πολλά έργα τα οποία υλοποιήθηκαν με την βοήθεια τη ΕΤΕΠ. Και υπήρχαν έργα τα οποία πήγαιναν πάρα πολύ καλά και πράγματα τα οποία γίνανε πάρα πολύ καλά, αλλά υπήρχαν και πολλά που θα μπορούσαν να βελτιωθούν. Η γραφειοκρατία, για παράδειγμα. Δεν καταφέραμε πάντα να πάρουμε ε, τα χρήματα όπως περιμέναμε από την ΤΕΠ. Μερικές φορές παίρναμε ε, περισσότερα, άλλες φορές έπρεπε να υπάρχει βελτίωση. Και πάρα πολλές φορές, υπερβολικά πολλές θα έλεγα, εάν τα έργα αυτά ήταν για ένα μείγμα πρωτοβουλειών για σύνολο ε, ιδιωτικών επενδύσεων μέσω ενδιάμεσων τραπεζών. Στο τέλος, οι τράπεζες αποφάσισαν για τη χρηματοδότηση της οικονομίας σαν να επρόκειτο για ιδιωτικές επενδύσεις καθαρά. Δηλαδή ο ρόλος της ΕΤΕΠ δεν ήταν ξεκάθαρος στα έργα αυτά, ούτε ο ρόλος των εθνικών αρχών. Ποια είναι η διαφορά από το αν έχουμε ιδιωτική τράπεζα ή όχι. Αυτό δεν ήταν σαφές. Χρειάζεται λοιπόν μεγαλύτερη εξασφάλιση και χρειάζεται μεγαλύτερο μείγμα στις πολιτικές μας. Χρειάζεται χρήμα και από τα κράτη, ίσως και από τη συνοχή, να μπουν μαζί με τα χρήματα της ΕΤΕΠ και έτσι να είμαστε σίγουροι ότι στηρίζουμε τα πιο ευάλωτα ε, προγράμματα και έργα. Το θέμα του άνθρακα και η μετάβαση στις πιο φτωχές περιοχές ε, θα είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Καταλαβαίνετε ότι οι βιομηχανοποιημένες περιοχές έχουν πολλές δυνατότητες, ενώ οι φτωχές περιοχές που χρειάζονται τη μετάβαση έχουν ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες να βρουν χρήματα από τράπεζες. Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε ε, δημόσιες πολιτικές και θα είναι πιο δύσκολο ε, για σας και το κράτος να στηρίξουν τέτοιου είδους έργα. Πάντω εμεί, την ΕΤΕΠ θέλουμε όταν λέει «Ε, θα γίνουμε πιο πράσινοι, ναι, αλλά με κόκκινη καρδιά. Δηλαδή θα πρέπει να δώσετε προτεραιότητα στις περιφέρειες και στις περιοχές εκείνες που είναι περισσότερο ευάλωτες και κινδυνεύουν περισσότερο από αυτή τη μετάβαση. Για εξού και ερώτησή μου, είσαστε έτοιμοι να δώσετε στήριξη με διαφορετικά μέσα και εργαλεία ε, που θα τα προσθέσετε στα χρήματα που δίνει το κράτος ή τα κονδύλια της συνοχής για να στηρίξετε τα πιο επικίνδυνα ε, προγράμματα στις περιφέρειες εκείνες που τα χρειάζονται. Χρειάζεται διαφοροποίηση λοιπόν. Και τέλος, ποια είναι η γνώμη σας, η προσωπική αλλά και της ΕΤΕΠ, για τον χρυσό κανόνα όσον αφορά τις δημόσιες επενδύσεις. Δεν είχαμε αρκετές δημόσιες επενδύσεις πρόσφατο, όπως ξέρετε. Δεν μπορέσαμε καν να επιστρέψουμε στα επίπεδα δημοσίων επενδύσεων που είχαμε πριν από την κρίση. Χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερες δημόσιες επενδύσεις εξού και στηρίζουμε την ιδέα ενός χρυσού κανόνα για τις δημόσιες επενδύσεις και κυρίως για πράσινες επενδύσεις. Χρειαζόμαστε αυτή την ευελιξία στους δημοσιονομικούς κανόνες για να προωθήσουμε περισσότερες επενδύσεις. Μπορείτε να μου πείτε αν συμφωνείτε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. η απάντηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα σχόλια που ήταν εφορτισμένα, έτσι, αλλά και για την ε, στήριξή σας στα διάφορα μέτρα. Πραγματικά μπορώ να πω ότι πράγματι αυτή είναι μια στιγμή που πρέπει να είμαστε εμεί προορατικοί, αλλά και να αντιδράμε στις διάφορες αλλαγές και να λάβουμε υπόψη μας όλες τις περιπτώσεις, τα δημοσιονομικά ιδρύματα, τις ε, αναπτυξιακές τράπεζες κλπ. και να μπορέσουμε όλα αυτά να τα συνδυάσουμε, να υπάρχει συνεργασία μεταξύ τους και να είμαστε έτοιμοι όντως να επενδύσουμε σε πιο, σε λιγότερο σίγουρα και ασφαλή έργα. Σίγουρα χρειαζόμαστε περισσότερες δημόσιες επενδύσεις και ναι και περισσότερη ευελιξία χρειάζεται όσον αφορά του δημοσιονομικού κανόνε, ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να ε, προχωρήσουν σε τέτοιου είδου έργα. Αλλιώ, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι για τις εθνικές κυβερνήσεις να κάνουν περισσότερες δημόσιες επενδύσεις εάν είχαν ε, πάρα πολύ αυστηρούς δημοσιονομικούς κανόνες. Δεν πρέπει βέβαια να πάμε στα άκρα. Θα είμαστε προσεκτικοί. Να μην πηγαίνουμε από το ένα άκρο στο άλλο. Μην πηγαίνουμε και σε υπερβολικά ανασφαλή έργα. Τώρα όσον αφορά την τράπεζα. Λέτε, αν είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε ε, μεγαλύτερο blending, μείγμα ναι, βεβαίως. Αυτή είναι η ιδέα πίσω από τον μηχανισμό της δίκαια μετάβασης και, και την τράπεζά μας. Ακριβώς αυτό θέλουμε να κάνουμε. Πέρα από τους μεταβατικούς μηχανισμούς, εμείς να δίνουμε επιπλέον χρήματα που εμείς κερδίζουμε από τις αγορές, να τα προσθέσουμε στα κονδύλια τα οποία ήδη προβλέπονται στον μηχανισμό δίκαιας μετάβασης. Περί αυτού πρόκειται κινητοποίηση κονδυλίων, μεγαλύτερο blending, μίξη επενδύσεων και κονδυλίων και μείγμα παντός χρηματοδότησης. Είπατε ότι ναι, τα πράγματα αλλάζουν στην αγορά σε σχέση με την περίοδο της κρίσης. Έχουμε περισσότερα χρήματα στις ε, κεφαλαγορές και έτσι μπορεί να υπάρξει κινητοποίηση και να έχουμε μεγαλύτερη μόχλευση και άρα μεγαλύτερη χρηματοδότηση. Οπότε, πραγματικά, υπάρχει χρηματοδότηση της ΕΤΕΠ, δημόσια, χρηματοδότηση, ιδιωτική χρηματοδότηση και επιπλέον από την Κομισιό. Νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να έχουμε περισσότερα χρήματα για επενδύσεις. Γιατί, όπως είπα, επιτρέψτε μου, έχουμε ένα μπουκέ, ένα μείγμα, ένα πακέτο με πολλά είδη χρηματοδότησης. Δίνουμε σημασία στην κοινωνική διάσταση, έτσι, με τη χρηματοδότησή μας και σίγουρα εκεί χρειάζεται, χρειάζονται επιχορηγήσεις, χρειάζονται και δημόσιες επενδύσεις με ανανέωση των τρόπων χρηματοδότησης και επενδύσεων ώστε να υπάρξει αναβάθμιση και στις δημόσιες υποδομές, αλλά χρειάζεται και τεράστια επένδυση από πλευρά του ιδιωτικού τομέα, ώστε να πετύχουμε αυτή τη νέα μετάβαση με τις ανανόσιμες πηγές, εναλλακτικέ πηγές ενέργειας και μέτρα ενεργειακής ε, ε, απόδοσης. Και μόνο με μείγμα επενδύσεων, μόνο με όλα αυτά τα είδη χρηματοδότησης μπορούμε να πετύχουμε. Περί αυτού πρόκειται. Αυτή είναι η μετάβαση. Και επίσης με το ταμείο της ΕΤΕ που θα κινητοποιηθεί επίσης, νομίζω ότι θα καταφέρουμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Από την ομάδα Renew, ο κύριος Μπιζού. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα σας κυρία Αντιπρόεδρε ε, και σας ευχαριστώ. Εδώ η Επιτροπή μας λέγεται Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικές είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, για τις περιφέρειές μας. Και ε, όλοι γνωρίζουν επίσης πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν μικρομεσαίες στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Είναι κεφαλαιόδου σημασία σε εργαλεία οι εταιρείε αυτές στην καταπολέμηση της ανεργίας. Αυτό ο ρόλος συνοχής, ο οικονομικός και ο κοινωνικός ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι ακόμα πιο σημαντικός στις πιο απομακρυσμένες και πιο ευαίσθητε και εύθραυστε περιφέρειες και σε ε, τις δικές μας περιφέρειες και ιδιαίτερα στις ε, άκρως απομακρυσμένες. Υπάρχει θέληση, υπάρχει ταλέντο, υπάρχουν ικανότητες και οι τράπεζες υπάρχουν. Θέλει ο κόσμος να επιχειρεί, αλλά οι τράπεζες ε, διστάζουν όλο και περισσότερο και δεν θέλουν να το ρισκάρουν. Είναι δουλειά τους να συνοδεύουν, να πλαισιώνουν και να ε, δίνουν αξία ε, στις επενδύσεις θα πρέπει γρήγορα να βρεθούν λύσεις ακριβώς για να αξιοποιηθούν και να βοηθηθούν όσοι άνθρωποι θέλουν να δημιουργήσουν και να δημιουργήσουν και θέσεις εργασίας. Επίγει αυτό από κοινωνική άποψη και είναι και μια άσκηση συλλογική ευφυία. Ευχαριστώ πολύ. Απάντηση. Κυρία Παύλοβα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μπιζού. Είναι πολύ σημαντική η ερώτησή σας και έχετε δίκιο. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Εκείνες χρειάζονται ακριβώς την υποστήριξη για την καινοτομία τους, δημιουργία θέσεων εργασίας, μέτρα ενεργειακής απόδοσης και οτιδήποτε χρειάζονται ιδιαίτερα σε αυτούς τους καιρούς μεταβατικούς. Είναι προτεραιότητα οι μικρομεσαίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ε, τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα χρηματοδοτικά μέσα που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Οι λεγόμενες πρωτοβουλίες για τις μικρομεσαίες. Εμείς τις υποστηρίζουμε. Και σε αυτή την προγραμματική περίοδο έχουν δώσει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα στην στήριξη των μικρομεσαίων. Όχι μόνο τις νεοφύς ε, επιχειρήσεις, αλλά και άλλες επιχειρήσεις υποστηρίζουμε καινοτόμες, τα μέτρα για την ενέργεια, την ενεργειακή απόδοση κτλ. Εκεί θα πρέπει να επικεντρωθούμε και να εστιάσουμε. Ιδιαίτερα στο δεύτερο πυλώνα πιστεύω, στο Invest in You. Έχουμε τις τέσσερις θηρίδες εκεί και τις διάφορες προτεραιότητες από τη μια και από την άλλη θα υπάρχει δυνατότητα αυτής της κάθετης προτεραιότητας ή ιεράρχησης για τα πράσινα έργα. Θα έχουμε λοιπόν έτσι μια καταπληκτική ευκαιρία να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες από το δεύτερο πυλώνα του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης και αυτό θα μας επιτρέψει ακριβώς να βοηθήσουμε περισσότερες. Τώρα στο σχέδιο Juncker έχουμε χρηματοδοτήσει ε, ένα εκατομμύριο μικρομεσαίες και φυσικά στις ε, άκρως απομακρυσμένες περιφέρειες, εξόχως απομακρυσμένες όπως λέγονται. Έχουμε παρατηρήσει κάποια διστακτικότητα, αλλά ποιος είναι ο δικός μας ρόλος. Εμείς δίνουμε εγγύηση ως τράπεζα. στις εγχώριες τράπεζες. Με τις δικές μας εγγυήσεις μπορούν οι εμπορικές τράπεζες, ε, οι εγχώριες να βοηθήσουν. Ε, ε, θα, υπό την προστασία την, την ομπρέλα, όπως το ονομάζουμε, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, μπορούμε να τις ενθαρρύνουμε να χορηγούν φθηνότερο χρήμα, μου επιτρέπεται, στις χώρες εκεί μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εξόχως απομακρυσμένες περιφέρειες. Μερικά στοιχεία αν θέλετε να σας δώσω. Γύρω στα 20 δις ήταν ο δανεισμός μας ε, μέσω κάποιων ενδιαμέσων. Χρησιμοποιούμε ε, τις ε, εκεί τράπεζες για να δανειδοτούμε τις επιχειρήσεις. Είναι από τα βασικότερα προϊόντα μας αυτά και συνεργαζόμαστε πραγματικά με πολλές εμπορικές τράπεζες ε, και στις εξόχως απόμακρες περιφέρειες θα πρέπει να το συνεχίσουμε αυτό, να το μεταξελίξουμε, γιατί θα πρέπει όλες οι περιφέρειες να ενισχύονται και να μην ε, μείνει κανείς παραπονεμένος. Ευχαριστώ. Ε, πρόεδρος, ευχαριστώ. Από την ομάδα ε, Ταυτότητα και Δημοκρατία, η Φραντσέσκα Ντονάτο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και σας κυρία Παύλοβα για αυτή τη σημαντική ανταλλαγή απόψεων. Καλύφθηκαν πολλές από τις ερωτήσεις μου, τις απαντήσεις που δώσατε ε, στους συναδέλφους. Συμφωνώ και συμμερίζομαι και εγώ τις ανησυχίες και τις αγωνίες των συναδέλφων ε, και τα όσα ρώτησα σε σχέση με αυτά που είπατε επιτρέψτε μου να πω κάποια πράγματα για τα όσα άκουσα από σας. Το σημαντικότερο από αυτά που είπατε ήταν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα είναι η έλλειψη επενδύσεων, η υποεπενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο ρόλος της ΕΤΕΠ είναι πρωταγωνιστικός για την προσέγγιση επενδύσεων, την ενθάρρυνση. Όπως είπατε όμως, αυτό που έχει σήμερα θεμελιώδη σημασία είναι να τονωθούν οι δημόσιες επενδύσεις. Και το ανέφεραν και οι συνάδελφοί μου, πολύ σημαντικά όλα αυτά τα θέματα. Για παράδειγμα, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης είναι κάτι που αξίζει την προσοχή μας θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να αποφύγουμε όλες οι επενδύσεις από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης να στραφούν ε, προς ε, τον άνθρακα και συναφείς ε, πηγές ενέργειας. Μάλλον να φύγουν από εκεί και να πάνε στις ανανεώσιμες. Γιατί υπάρχουν και άλλοι τρόποι να έχεις μια κυκλική οικονομία και νέες πηγές ενέργειας ε, που χρειάζονται και αυτές χρηματοδότηση. Υπάρχουν πολλές ευρωπαϊκές περιφέρειες που μπορούν κατά αυτόν τον τρόπο να γνωρίσουν μία βιώσιμη ανάπτυξη. Θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα εφαρμοστούν τα κριτήρια αυτά. Προτείνω ευελιξία όσο περισσότερο γίνεται, έτσι ώστε να μπορέσουν όλες οι χώρες να υποφεληθούν και να έχουν πρόσβαση στα κονδύλια αυτά και στην χρηματοδοτική ε, υποστήριξη. Συμφωνώ επίσης με τη σημασία που πρέπει να δοθεί στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα των μικρών. Έχει πάρα πολύ μεγάλο δίκιο ο συνάδελφος. Υπάρχουν πολλές ε, περιφέρειες απομακρυσμένες ε, ε, στην περιφέρεια της Ευρώπης ακριβώς και είναι πάρα πολύ δύσκολο οι μικρές επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση ε, στην δανειοδότηση από τις τράπεζες. Και είναι σημαντικό τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως το δικό σας, να βρουν έναν τρόπο να φτάνουν μέχρι αυτές τις μικρές επιχειρήσεις. γιατί η έλλειψη αυτής της υποστήριξης είναι από τους βασικότερους λόγους για τους οποίους εμφανίζουν καθυστέρηση κάποιες περιφέρειες. Είναι και ο ιστό ε, της οικονομίας μας ε, που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή μεγάλες δυσκολίες. Και θα πρέπει να υποστηριχθούν οπωσδήποτε οι μικρές επιχειρήσεις. Με οποιοδήποτε τρόπο. και με νομοθετικές παρεμβάσεις ενδεχομένω από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, έτσι ώστε η τοπική αυτοδιοίκηση να μην πώς να το χρησιμοποιεί αθέμητες μεθόδους για να σταματήσει τις επενδύσεις. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Καμιά φορά οι τοπικές αρχές και η αυτοδιοίκηση ε, χρησιμοποιούν ως πρόφαση, πώς να το πω τώρα στα αγγλικά, Ε, την ακαιρεότητα του τοπίου και τη διαφύλαξη του τοπίου για να σταματήσουν επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά, Φερρυπίν. Θα πρέπει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να επεμβαίνουν για να μην μπορούν να εμποδίζουν την ανάπτυξη οι τοπικές αρχές και να προχωρήσουμε στην κυκλική οικονομία και στην πράσινη οικονομία. Εν πάση περιπτώσει, εγώ σας εμπιστεύομαι ότι θα κάνετε ό,τι μπορείτε προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ. Θα σας αφήσω να απαντήσετε παρόλο που κανονικά θα έπρεπε να δώσω το λόγο στη συνάδελφο για τους πράσινους, αλλά αμέσως μετά απαντήσετε θα λάβουν το λόγο. Παρακαλώ λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Αντωνάτο οι υποεπενδύσεις είναι ένα πραγματικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε και θα πρέπει να κινητοποιήσουμε όλα τα όργανα ε, και να κινητοποιηθούμε για να βρούμε μια λύση. Έχουμε όμω το μηχανισμό που προτάθηκε και με όλες τις προσπάθειες που έχουμε κάνει και τις άλλες πηγές χρηματοδότησης πιστεύω πως είμαστε σε σωστή τροχιά. Και θέλω να επαναλάβω, μια και έχω την ευκαιρία, πως αν εξετάσουμε τους τρεις άξονες του Μηχανισμού για τη Δίκαιη Μετάβαση. Συνολικά και σφαιρικά αντιμετωπίζουμε το θέμα. Ο πρώτος πυλώνας είναι η κοινή διαχείριση στα, που βασίζεται στα επιχειρησιακά προγράμματα και στις περιοχές συνοχής και στη συμπληρωματικότητα με τις επενδύσεις. Ο δεύτερος πυλώνας έχει να κάνει με τη στήριξη, τη πραγματική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των βιομηχανιών και σε όσους χρειάζονται να κάνουν αφενός μία μετάβαση και αφετέρου να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί και να αναπτυχθούν. Και ο τρίτος πυλώνας είναι η οικονομική αναγέννηση που εστιάζεται κυρίως, όπως το ονομάζουμε εμείς, γιατί είναι ουσιαστικά εκεί που ε, οι κανόνες οι δικοί μας ε, αποφασίζουν. Ο τρίτος πυλώνας λοιπόν είναι η δυνατότητα που έχουμε να χορηγήσουμε ε, δάνεια στο δημόσιο τομέα για να τον στηρίξουμε για όλη την επταετία για να μοχλεύσει 25 με 30 δις επενδύσεων με χορηγίες, με επιδοτήσεις σε έργα που είναι υποδομές ε, ενέργειας, μεταφορών, τηλεθέρμανση, ΑΠΕ Όλα αυτά όμως ε, από την πλευρά του δημοσίου. Και αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο έχει ε, κατανεμηθεί το Ταμείο για τη Δίκαια Μετάβαση. Άρα λοιπόν στο δημόσιο κλάδο εμείς εκεί μέσω του τρίτου πυλώνα θα στηρίξουμε με τις απαραίτητες επενδύσεις και τα δικά μας ε, χρηματοδοτικά εργαλεία. Και νομίζω ότι αυτή είναι και μια καλή ευκαιρία για μας να κάνουμε κάτι παραπάνω εκεί. Βεβαίως και, στη δεύτερη, ε, και στο δεύτερο πυλώνα στηρίζουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν έχουμε ένα διτό ρόλο, δεύτερος και τρίτος πυλώνας, μικρομεσαίες και δημόσιος κλάδος και έχουμε εμπειρία και στα δύο και πιστεύω πως θα πρέπει να ε, στηρίζουμε βήμα-βήμα και για να πετύχουμε χρειάζεται και μία θετική ε, εθνική συμμετοχή που θα έχει τη μορφή των εθνικών στρατηγικών. Γιατί θα πρέπει να αξιολογήσουμε συγκεκριμένα τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά κάθε διαφορετικής περιφέρειας. Γιατί κάθε μία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Και θα πρέπει να τα βρούμε, να τα λάβουμε υπόψη και βέβαια θα πρέπει κάθε κράτος μέλος να ε, προ η μέτρα, να εντοπίσει αυτές τις περιφέρειες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, να το στηρίξουμε μέσω της δικής μας συμβουλευτικής ε, και των ε, εμπειρογνώμων μας. Αλλά τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ξεκινήσουν με προτάσεις, τις οποίες θα συμφωνήσουν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά να στηρίξουμε εμείς. Ευχαριστώ πολύ. Κλασνίνας από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Η πρώτη μου ερώτηση είναι εξής. Έχουμε ακούσει τόσα πολλά για την απόφαση της ΕΤΕΠ να γίνει πράσινη, να γίνει κλιματική τράπεζα και για να μην αναφέρω όσα ακούγονται ότι μπορεί να πρόκειται για μια πολιτική που τελικά κατευθύνεται από την ιδεολογία. Εγώ θα αναφερθώ περισσότερο στους οικονομικούς λόγους που κρύβονται πίσω από την απόφαση αυτή. Γιατί έχουμε δει ότι το ρηκτά, τα πυρηνικά δεν φτάνουν. Δημιουργούν οικονομική αβεβαιότητα και ότι πολλοί επενδυτές απομακρύνονται από αυτά. Ε, κάποιο, ο κ. Μπάφετ, ίσω να τον έχετε ακούσει, είναι ο μεγαλύτερο επενδυτή στον κόσμο. Εγώ δεν συμφωνώ βέβαια καθόλου με τι επενδύσει του, αλλά αποφάσισε να απομακρυνθεί από παντός είδου ε, καύση ορυκτών γιατί πιστεύει ότι δεν έχουν μέλλον οι επενδύσεις του εκεί. Οπότε εγώ θέλω να ξέρω ποιοι είναι οι οικονομικοί λόγοι που σας απομακρύνουν από τα ορυκτά και από την στήριξη πυρηνικών ή Και κάτι ακόμα. Αναφερθήκατε στις εθνικές στρατηγικές για το μηχανισμό δίκαιας μετάβασης. Πιο συγκεκριμένα, τι περιμένετε από τις χώρες μέλη να κάνουν και πώς εσείς βοηθάτε ώστε να προχωρήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση οι μέλη, ώστε οι δικές τους στρατηγικές ευθυγραμμίζονται με την πραγματικότητα των αναγκών για την μετάβασή του. Και τι γίνεται με παλιά σχέδια επενδύσεων που υπάρχουν από το παρελθόν και τώρα με την ε, νέα πράσινη συμφωνία αλλάζει η κατάσταση. Οι παλιές ιδέες επενδύσεων του παρελθόντος δηλαδή που πήγαιναν σε ένα μεγάλο βαθμό ε, στην καύση ορυκτών. Πιστεύετε ότι αυτό θα επηρεάσει τα στρατηγικά σχέδια και τι θα κάνει η ΕΤΕΠ και πώς θα στηρίξει τις χώρες μέλη ώστε να καταλήξουν στη σωστή ε, απόφαση όσον αφορά τις δικές τους επενδύσεις. Απάντηση. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Πολλές σοβαρές ερωτήσεις. Και εδώ δεν πρόκειται μόνο για την ΕΤΕΠ, πρόκειται και για τον ίδιο το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί όπως γνωρίζετε, είναι πρώτα οι χώρες μέλη που πρέπει να σχεδιάσουν τα δικά του σχέδια μετάβασης, που θα καθοριστούν από τις χώρες μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Φυσικά, έχοντας υπόψη την κατάσταση, εμείς Βεβαίω και είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε κατευθυντήριε γραμμέ και στήριξη με την συμβουλευτική μα ομάδα, να στηρίξουμε την εκπόνηση στρατηγικών καταρχήν και σε ένα μετέπειτα στάδιο την ε, παραπέρα ανάπτυξη της ε, πρότασης για αναπτυξιακά έργα. Πάντως, τα αρχικά βήματα γίνονται στις χώρες μέλη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι δικός τους ρόλος να εντοπίσουν που θέλουν να επενδύσουν και να αποφασίσουν για τις πολιτικές τους. Δεν εκπονούμε εμείς πολιτική. Και μετά, βεβαίω όπου μπορούμε και εμείς, ε, βοηθάμε, στηρίζουμε. Υπάρχουν ε, διαφορετικοί τρόποι γι' αυτό. Σας είπα ότι μπορούμε να βοηθήσουμε συμβουλευτικά αφενός και με δανεισμό αφετέρου. Τώρα το είπα και πριν στην προηγούμενη ερώτηση, αλλά το ξαναλέω. Έχουμε ένα συγκεκριμένο καταστατικό που δεν μας επιτρέπει να βάζουμε κριτήρια ε, για χώρες ή για περιφέρειες, δηλαδή να είναι ανάλογα με τη χώρα ή ανάλογα με την περιφέρεια. Όχι. Είναι τραπεζικά τα κριτήρια επιλεξιμότητας και βεβαίως να υπάρχει δέος επιμέλεια. Και βοηθάμε για να προετοιμαστεί καλύτερα το σχέδιο, να μπορεί να χρηματοδοτηθεί τραπεζικά περνάει από την ε, χρηστική μας επιτροπή, από τις διάφορες διαδικασίες στην τράπεζα. Είμαστε μια τράπεζα, έτσι. Και ακολουθούμε όλα τα βήματα που ακολουθεί μια τράπεζα. Και μια που μιλάμε για την επιλεξιμότητα και τα κριτήρια αυτά, γίνονται συζητήσεις στην τράπεζα. Και υπήρξε κάτι που υιοθετήσαμε, που είναι μια νέα στρατηγική δανεισμού για την ενέργεια, το Δεκέμβριο εγκρίθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο με 94% των ψήφων, που σημαίνει με πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Και η απόφαση ήταν ότι δεν θα χρηματοδοτεί πια η τράπεζά μας από το τέλος του 2021 έργα που βασίζονται στον άνθρακα. Έτσι κι αλλιώς όλο και λιγότερο, αλλά σίγουρα από το τέλος του 2021 δεν θα υπάρχει πια τέτοια χρηματοδότηση. Όμως υιοθετήσαμε και νέα κριτήρια εκπομπών για τα νέα έργα που θα χρηματοδοτήσουμε στο μέλλον. Πριν είμαστε στο 550, τώρα είμαστε πολύ πιο χαμηλά. Έτσι λοιπόν η νέα ενεργειακή μας, ε, η νέα πολιτική μας για δανεισμό στα θέματα της ενέργειας όντως αλλάζει. Αυτές είναι οι αρχές πάνω στις οποίες ε, βασιζόμαστε εφ' για τον δανεισμό μας. Ενεργειακή απόδοση είναι το ένα, με νέους στόχους που συμφωνήθηκαν στην οδηγία για την ενεργειακή απόδοση έπειτα για αποφυγή άνθρακα υπέρ των τεχνολογιών μηδενικού άνθρακα μέχρι το 2030 και το τρίτο είναι ότι αυξάνουμε την χρηματοδότηση για καινοτόμες μορφές αποθήκευσης, ε, την ε, κινητικότητα και πράσινες επενδύσεις. Είμαστε υπέρ των ελλακτικών πηγών, ηλιακής, αιωλικής και στηρίζουμε βέβαια και την ενεργειακή ε, τροποποίηση. Για τέτοιου είδου έργα που καλύπτονται από την ε, πολιτική μας, θα χρηματοδοτούμε με 75%, όχι με 50% όπως κάνουμε για τα υπόλοιπα. Μέχρι 75% για να επωφεληθούν όσοι μπορούν από τον εξυγχρονισμό αυτόν τον ενεργειακό. Έτσι λειτουργούμε και έτσι έχουν οι κανόνες μας επιλεξιμότητας. Στο μεταξύ πάντως τώρα προχωρούμε και σε κριτήρια επιλεξιμότητα σε βάση συμμόρφωση στη Συμφωνία του Παρισιού. Τον Απρίλιο θα έχουμε καταλήξει σε αυτό. Και ετοιμάζουμε και έναν χάρτη πορείας τραπεζικό για να δούμε πώς εμείς θα προχωρήσουμε με τις φιλοδοξίες μας ε, βάσει του πεντετούς κύκλου που ακολουθούμε και ευχαρίστως όταν ε, έχει υιοθετηθεί αυτό το νέο κριτήριο, ευχαρίστως να έρθω και να σας το εξηγήσω τον Απρίλιο, τον Μάιο, φέτος. Έτσι θα έχουμε προχωρήσει, θα έχουμε κάνει άλλο ένα βήμα ε, προς τους στόχους μας. Έπειτα υπάρχει και το θέμα των μεταφορών και του δανεισμού μας στις μεταφορές και αυτό θα επανεξεταστεί η πολιτική δανεισμού μας δηλαδή στις μεταφορές, το δεύτερο εξάμεινο φέτος. Περιμένουμε όμως την αναθεώρηση της στρατηγικής από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα γίνει το Σεπτέμβριο. Οπότε μετά θα γίνει διαβούλευση, δημοσία συζήτηση και εδώ ευχαρίστω να έρθω και να το συζητήσω και μαζί σας στην Επιτροπή αυτή. Γιατί πιστεύω ότι ο δανεισμός στις μεταφορές είναι ένα σημαντικό τμήμα των υποδομών και όχι μόνο των υποδομών. Πρέπει να στηριχθούν οι μεταφορές στο μέλλον. Η πολιτική μας μεταφορών δεν έχει προσαρμοστεί από το 2011 και μετά. Τώρα έχουμε νέους στόχους να πετύχουμε. Συνεπώς, αυτή είναι άλλη μια πρόκληση που μας περιμένει όσον αφορά τα πυρηνικά. Δεν αποτελεί μέρος της δικιάς μας πολιτικής δανεισμού. Δεν χρηματοδοτούμε νέες πυρηνικές μονάδες. Το μόνο που ίσως χρηματοδοτήσουμε στην μεταβατική περίοδο είναι μέτρα ασφάλειας για πυρηνικούς σταθμούς που ήδη υπάρχουν όμως, όχι για νέους. Υποδομές και τέτοια όχι καθόλου. Αυτή είναι η κατάσταση. Μπορώ να σας δώσω και περισσότερες λεπτομέρειες αν θέλετε, αλλά Εντάξει, θα σταματήσω εδώ προς το παρόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σπυράκη, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Κυρία Παύλοβα, σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε σήμερα στην Επιτροπή μας για να συζητήσουμε ζητήματα που άπτονται της Πράσινης Συμφωνίας και του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης. Όπως γνωρίζετε, στην Ελλάδα έχουμε την περιοχή, την περιφέρεια της Δυτικής ε, Μακεδονίας και μια άλλη πόλη που είναι η μεγαλόπολη στη Πελοπόννησο που εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον άνθρακα. Για να καταλάβω τι πρέπει να κάνουμε. Αρχίζω από το ποσοστό συνεισφοράς ε, της ΕΤΕΠ ε, στο Invest EU. Ποιο θα είναι το ποσοστό της δικής σας χρηματοδότησης και τι θα μοχλεύσει. Ποια θα είναι η διαδικασία μόχλευσης. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι έτοιμη να αρχίσει να συνεννοείται με τον κόσμο επιτόπου. Γιατί υπάρχει μια τράπεζα εκεί που εξετάζει το σχέδιο, αλλά η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει σημασία να έχει παρουσία επιτόπου, γιατί εκκρεμούν πολλά ζητήματα. Ας πούμε τι γίνεται με τον ενεργειακό ανεφοδιασμό για την τηλεθερμία, ε, τηλεθέρμανση στη Δυτική Μακεδονία. Το φυσικό αέριο θα το χρηματοδοτήσατε, είπατε, μέχρι το 2021. Αλλιώς θα πρέπει να προέρχεται η χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για να ολοκληρωθεί το έργο. Και ένα τρίτο είναι ο τρόπος που θα δοθεί η τεχνική ε, βοήθεια Πώς θα συνεννοήσετε εκεί με την τοπική αυτοδιοίκηση ή θέλετε να παραμείνετε σε διεθνές επίπεδο και να υποστηρίζετε τη διαδικασία μέσω των εθνικών σχεδίων για την μετάβαση. Ευχαριστώ πολύ. Απάντηση. Κυρία Αντιπρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Όντως, πολλές περιφέρειες εξαρτώνται από τον άνθρακα. Και όπως είπα, το πιο σημαντικό για τις περιφέρειες αυτές είναι να χαράξουν μια περιφερειακή στρατηγική για τη μετάβαση με συγκεκριμένες στρατηγικές και βήματα για τη μετάβαση, έτσι ώστε να εξηγηθεί πώς θα γίνει αυτή και τη χρονική της διάρκεια. Είναι μία προσέγγιση από την βάση προς την κορυφή, είναι απαραίτητο αυτό και σίγουρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα σας στηρίξει για να αναπτύξετε αυτή την ε, στρατηγική. Αν θεωρηθεί απαραίτητο, η δική μας ε, ομάδα συμβούλων θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει, να στηρίξει στην περιφέρεια αυτή γιατί εμείς δεν στηρίζουμε μόνο κεντρικές κυβερνήσεις, αλλά επίσης και τοπικές, την τοπική αυτοδιοίκηση. Οπότε με χαρά σας παρουσιάσω τους ε, συναδέλφους μου από τη μονάδα ε, παροχής συμβουλών κτλ. Οπότε μπορούμε να σας δώσουμε περισσότερες προφορίες για το πώς λειτουργούν όλα αυτά. Για να συνεισφέρουμε περισσότερο. Μέσω ε, τεχνικών συμβουλών. Τώρα για τους ίδιους τους πυλώνες που ρωτήσατε πώς γίνεται η μόχλευση. Όπως σας είπα, με τον πρώτο πυλώνα δεν έχουμε καμία σχέση. Έχουμε ρόλο ε, στον πυλώνα 2 και στον πυλώνα 3. Στο δεύτερο πυλώνα 1,8 δις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο δεύτερο πυλώνα ως εγγύηση και με την εγγύηση αυτή και με τους ίδιους πόρους που έχουμε εμείς ως ΕΤΕ, θα μοχλεύσουμε μέχρι 45 δις ευρώ επενδύσεων. Δηλαδή, Το δικό μας μερίδιο από την ΕΤΕ είναι γύρω στα 10-15 δις, έτσι ώστε να έχουμε αυτό τον παράγοντα μόχλευσης, ο οποίος ε, έτσι θα λειτουργήσει. Για τον τρίτο πυλώνα, που έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση του δημοσίου τομέα, είναι ένας μηχανισμός ο οποίος έχει ε, και ένα σκέλος που είναι οι ε, ενισχύσεις, η χορήγηση ενισχύσεων και είναι η ενεργειακή ε, αποδοτικότητα, η ενεργειακή αναβάθμιση ή τηλεθέρμανση, όντως, με καινοτόμες λύσεις. Και εκεί το πιο σημαντικό που θα πρέπει να κρατήσετε είναι πως εμείς στηρίζουμε τα έργα τα οποία δεν παράγουν ε, αρκετά έσοδα έτσι ώστε να μπορούν να αυτοχρηματοδοτηθούν. Αν λοιπόν ένα έργο δεν μπορεί ε, να χρηματοδοτηθεί ε, μέσω μιας εμπορικής τράπεζας γιατί δεν παράγει έσοδα, μπορείτε να μας ζητήσετε να συνεισφέρουμε με επιπρόσθετη χρηματοδότηση για να λάβει σάρκα και οστά. και να προσφέρει με αποτελεσματικό τρόπο στην ίδια την περιφέρεια. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πασκάλα Ριμόντο, ευχαριστώ πολύ κυρία Παύλοβα. Τα τελευταία χρόνια έχω συναντηθεί αρκετές φορές με τα μέλη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και έχω καταλάβει πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της τράπεζας στην Ευρώπη. Τα επόμενα έτη μπορεί να κληθεί να διαδραματίσει διαφορετικό ρόλο η τράπεζα. Και έχω δύο ερωτήσεις εκεί. Η μία ερώτηση έχει να κάνει με τις ιδιωτικές επενδύσεις. Την περασμένη εβδομάδα και την προπερασμένη εβδομάδα ακούσαμε κάποια αριθμητικά στοιχεία που δείχνουν ότι θα έχουμε ε, πολλές ιδιωτικές επενδύσεις μετοχιακές ε, στην αηφόρο ανάπτυξη. Ας πούμε, ε, το είπαν και η πράσινη Ανέφερε ο συνάδελφος Νίνας ότι μέχρι και ο Warren Buffett αποφάσισε να μην επενδύει πια σε ορυκτά κάψιμα και να επενδύει μόνο σε μετοχές ε, βιώσιμης ανάπτυξης. Ερωτώ λοιπόν, τι ρόλο μπορεί να διαδραματίσει εκεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων όταν φτάσουν αυτά τα χρήματα στην αγορά και πέσουν σε επενδύσεις στην Ευρώπη. Ένας επενδυτής που επιθυμεί ε, να επενδύσει έστω και στη βιώσιμη οικονομία παραμένει επενδυτής και θέλει να έχει κάποιο κέρδος όταν επενδύει κάπου. Τι θα συμβουλεύει η τράπεζα στους πελάτες. Ε, ε, πάντα οι τράπεζες συμβουλεύουν επενδύσεις που αποφέρουν. έρχεται ας πούμε ένα ταμείο, ένα φαντ και θέλει να επενδύσει βιώσιμα στην Ευρώπη. Εσείς πού θα το προσανατολίσετε, σε ποια έργα θα το στρέψετε. Γιατί το αποφασιστικό επιχείρημα δεν είναι το βιώσιμο, είναι πόσο θα βγάλω εγώ ως επενδυτής. Και ένα δεύτερο λογιστικό. Είπατε ότι και στο μηχανισμό δίκαιης μετάβασης ή το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης υπάρχει ένας τρίτος πυλώνας ο οποίος έχει στόχο τις δημόσιες επενδύσεις ή να βοηθάει το δημόσιο να κάνει επενδύσεις σε έργα που έχουν νόημα. Το δημόσιο έχει ένα πρόβλημα γιατί έχει κάποια λογιστικά πρότυπα. Υπάρχει ένα πρότυπο που λέγεται SEC, ε, το οποίο είναι πρόβλημα ή υποχρέωση για το δημόσιο. Σε μία επένδυση, ας πούμε, όταν ε, υλοποιείτε το πρόγραμμα θα πρέπει να εγγράφετε λογιστικά εκείνο το έτος. Και ε, και δεν μπορεί το κράτος να το μοιράσει σε διάφορα χρόνια, όπως μπορεί μια ιδιωτική επιχείρηση, για να αποσβέσει ε, αυτή την δαπάνη. Και ε, αυτό είναι φρένο και τροχοπέδι για τα κράτη, γιατί κινδυνεύει να ξεφύγει το κράτος από τον ισοσκελισμένο προπολογισμό όταν εγγράψει σε ένα μόνο έτος μια τέτοια επένδυση. Ε, θέλει το δημόσιο να κάνει επενδύσεις, αλλά είναι δεμένα τα χέρια του από ε, τους ισχυρά άκαμπτους κανόνες τήρησης λογιστικών βιβλίων. Είναι αυτά τα πρότυπα ΣΕΚ για το δημόσιο Πώς μπορείτε να βοηθήσετε έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα με τους ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς των κρατών και να μην ξεφεύγουν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις αυτές, πολύ συγκεκριμένες. Ε, παρακαλώ, απαντήστε. Uh, thank you very much. Uh, to be really honest, I don't have all. Για να είμαι ειλικρινή, δεν έχω όλες τις απαντήσεις που χρειάζεται τώρα και συγκεκριμένα για ε, τα θέματα του offset και της λογιστικής ε, δεν μπορώ να απαντήσω παρά μόνο θα χρειαστεί ε, να δούμε τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τον αντιλογισμό και μετά θα σας απαντήσουν οι επαγγελματίες μια και είναι τεχνικά θέματα. Όντως, πάντως, με τις δημόσιες υπηρεσίες έχουμε αφενός το πρόβλημα του ελλείμματος όταν υπάρχουν τέτοιου είδους επενδύσεις και το δεύτερο ε, είναι ο λογιστικός αντιλογισμός. Οπότε θα πρέπει να το συζητήσουμε για να μπορέσω να σας δώσω μια πιο συγκεκριμένη απάντηση για τους βασικούς επενδυτές και για τη βιωσιμότητα και την κερδοφορία των επενδύσεων, νομίζω εκεί βρίσκεται ακριβώς και ο ρόλος μας. Εκεί καλείται να παίξει το μεγάλο ρόλο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και εμείς στην τράπεζα είμαστε πιο συντηρητικοί. Ε, δημιουργώντας λοιπόν αυτό το εργαλείο, αυτό το ταμείο, το ξεπερνάμε και έχω εδώ και τους συναδέλφους οι οποίοι μπορούν να σας δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες σε μια άλλη συνάντηση. Πάντως, τα εργαλεία και οι επενδύσεις που προτείνουμε μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε ε, περισσότερες ε, ε, επενδύσεις με κεφάλαια κινδύνου και μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους. Γιατί χωρίς τις ιδιωτικές επενδύσεις δεν θα καταφέρουμε ποτέ τίποτα. Αυτοί είναι οι ιδιώτες επενδυτές, οι μεγάλοι ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι αποτελούν και το στόχο μας. Τους χρειαζόμαστε. Χρειάζεται να τους προσελκύσουμε, χρειάζεται να επενδύσουν και παράλληλα εμείς είμαστε οι καταλήτες, το 1 τρίτο ε, των επενδύσεων γίνεται από το δικό μας όμιλο ε, τα υπόλοιπα προέρχονται είτε από τους μεγάλους επενδυτές, είτε από άλλες πηγές. Εμείς είμαστε, αν θέλετε, είμαστε συνυπενδυτές, αλλά παράλληλα είμαστε και σφραγίδα ποιότητας μιας επένδυσης. Δίνουμε το πράσινο φως, κάποιο είδους εξασφάλιση και ε, μιλάμε και για τη βιωσιμότητα του της επένδυσης την οποία εμείς κατά κάποιο τρόπο ε, εξασφαλίζουμε. Αυτό είναι το επιχειρηματικό μοντέλο και με τον τρόπο αυτό λειτουργεί. Και με τον τρόπο αυτό παραδίδει τα παραδοτέα τελικά. result oriented doing έτσι λοιπόν λειτουργεί η μόχλευση και πιστεύω ότι έχουμε καταφέρει καλά. Μάλιστα, καταφέραμε να μοχλεύσουμε λοιπόν αυτά τα 85 δις και να μεγιστοποιήσουμε τα αποτελέσματα, να φτάσουμε τα 460 δις συνολικά. Οπότε έχουμε αυτή την σφραγίδα ποιότητας που ε, προσφέρουμε. Παίρνουμε μια, αν θέλετε, δεύτερη θέση, αλλά ουσιαστικά ο ρόλος μας είναι τούτος. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Ο κύριος Όλμπριχτ. Ευχαριστώ πολύ. Τρεις ερωτήσεις έχω. Μία πολιτική και δύο τεχνικές. Ευχαριστώ που ήρθατε. Χαίρομαι που σας συναντάω και πάλι. Προσπαθώ λοιπόν να καταλαβαίνω τι ακριβώς εννοείται ότι θα γίνει η πράσινη τράπεζα, κλιματική τράπεζα, η ΕΤΕΠ. Τι ακριβώς εννοείται. Ακούγεται καλό, αλλά ακούγεται και κάπως μοδάτο. Σημαίνει κάτι σημαντικό όσον αφορά τη δομή. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Δεύτερον, κάτι που γίνεται όλο και πιο καυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι το θέμα αυτό της ταξινόμησης, δηλαδή πώς ταξινομούμε τις επενδύσεις σε επενδύσεις που ε, γίνονται για την προστασία του περιβάλλοντος ή όχι. Λοιπόν, ε, λέμε ότι θέλουμε να επιλέξουμε τις επενδύσεις ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα που θα γίνουν αποδεκτές από την ΕΤΕΠ εφόσον είναι προσανατολισμένες στην προστασία του περιβάλλοντος. Θέλω να μου το εξηγήσετε αυτό. Και τρίτον, είμαι λίγο, βλέπετε, βλέπω τα πράγματα κάπως ύποπτα. Γιατί ε, μας παρουσιάστηκαν πέρυσι νούμερα για συγκεκριμένες χώρες μέλη και εγώ είδα ποια είναι η κατανομή για τον πρώτο πυλώνα, 7,5 αν υπάρχουν χρήματα, αν δεχτούν τα κράτη-μέλη, θα είναι 7,5 και θα μοιραστούν στις 27 χώρες μέλη. Αλλά ε, στο, στα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουμε εκτιμήσεις για το δεύτερο και τον τρίτο πυλώνα. Μπορείτε λιγάκι να μας εξηγήσετε τι σημαίνουν αυτές οι εκτιμήσεις. Τι λένε δηλαδή ότι αν εργαστείτε πολύ καλά θα μπορέσετε να φτάσετε μέχρι. Γιατί το να κάνει κανείς εκτιμήσεις μπορεί το αποτέλεσμα να είναι πολύ ενδιαφέρον, όπω το ξέρετε. Εγώ ξέρω ότι βρίσκεται από πίσω, γιατί στη δικιά μου τη χώρα, για παράδειγμα, στην Πολωνία, η κυβέρνηση παρουσίασε τα πράγματα και είπε ότι έχει 30 δισεκατομμύρια συμπεριλαμβανομένων των εκτιμήσεων. Οπότε, εγώ θέλω να ξέρω στη συγκεκριμένη περίπτωση τι σημαίνουν οι εκτιμήσει για το δεύτερο και τον τρίτο πυλώνα. Για τον πρώτο το καταλαβαίνω, αλλά για το δεύτερο και τον τρίτο δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πολιτικό νόημα τη εκτίμηση. Ευχαριστούμε πολύ. Η Αντιπρόεδρος, παρακαλώ να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Όλμπρεχτ και εγώ χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Πράγματι έχετε δίκιο. Ξεκινάω λέγοντας και για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, όλες αυτές οι εκτιμήσεις βεβαίως είναι η πιο θετική περίπτωση, η πιο ευνοϊκή. Πρέπει όντως να κάνουμε προσπάθειες, να φροντίσουμε για τις αγορές μας, τον ιδιωτικό τομέα, την αγορά, με κάθε μέσο που διαθέτουμε, ώστε να κινητοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερα τα πράγματα για να φτάσουμε στον νότο επίπεδο γιατί όλοι οι στόχοι, οι φιλοδοξίες και τα λοιπά δεν είναι σίγουρα πράγματα. Έχουμε λοιπόν τα χρήματα που έχουμε και έχουμε και την, το αποτέλεσμα της κινητοποίησης που θα γίνει. Και πρέπει πράγματι να φροντίσουμε να δρομολογήσουμε όσο γίνεται ε, καλύτερα αποτελέσματα. Και αυτό θα γίνει με όσο γίνεται καλύτερη κινητοποίηση. Παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποια στοιχεία, αναχώρα με ποσοστά. Αλλά όπως είπα, είναι κάτι που εξελίσσεται. Πρόκειται για σχέδια προτάσεων έτσι κι αλλιώς, θα συζητηθούν ακόμα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις χώρες μέλη και μας τους ίδιους. Αν κοιτάξουμε τώρα, έτσι όπως έχουν οι δομές μας, δεν έχουμε ποσοστά για χώρες μέλη. Δεν έχουμε αυτή την προσέγγιση προς το παρόν. Προς το παρόν μπορεί να αλλάξει αυτό. Αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να αποφασίσει αν θα έχει κριτήρια για διαφορετικές χώρες ή για διαφορετικές περιφέρειες. Γιατί προς το παρόν το μόνο που μπορούμε να προτείνουμε είναι να στηρίξουμε όλες τις χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο να τις στηρίξουμε για τα έργα ώστε να μπορέσουν εκείνες να φτάσουν στο ανώτατο και να πετύχουν το στόχο με συμβουλές, με στήριξη, με κατευθυντήριες γραμμές, ίσως και με περισσότερα έργα, ώστε να υπάρχει κάλυψη και να υπάρχουν καλά έργα, τραπεζικά καλά έργα για τους διάφορους πυλώνες, κυρίως για τον τρία ώστε να επιτευχθεί ο στόχος. Αλλά αυτό είναι το μόνο που μπορούμε να προτείνουμε τώρα. Δεν μπορούμε, δεν δικαιούμαστε να κάνουμε κάτι άλλο. Αν αποφασίσει κάτι διαφορετικό το Διοικητικό Συμβούλιο, τότε μπορούμε να αλλάξουμε. Είμαστε ευέλικτοι. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει κάτι διαφορετικό, θα συμφωνήσουμε και θα καθορίσουμε κάποιες ποσοστώσεις αναχώρα. Το Διοικητικό Συμβούλιο όμως αποφασίζει. για την επιλογή των επενδύσεων υπέρ ε, της προστασίας του κλίματος και του περιβάλλοντος. Ναι, για να πετύχουμε τον ε, στόχο μας και για να έχουμε 50% του δανεισμού για κλιματικά προγράμματα, πράσινα κτλ. Ναι, πράγματι θα προσπαθήσουμε να ενθαρρύνουμε ώστε οι επενδύσεις μας να έχουν κλιματική διάσταση. Αλλά μην περιμένετε ότι όλα τα έργα θα έχουν 50%, ένα θα έχει 8%, ένα θα έχει 20% και μετά στο τέλος θα πρέπει να βγάλουμε το μεσόρο. Δεν θα επιμείνουμε κάθε έργο να έχει 50% ε, περιβαλλοντική διάσταση. Θα υπάρχει διαφοροποίηση. Άλλο έργο θα έχει μεγαλύτερη, άλλο μικρότερη διάσταση, εξαρτάται. για το τι σημαίνει στην πράξη η αλλαγή αυτή της τράπεζας σε κλιματική. Πολλά σημαίνει. Πρώτα απ' όλα, πώς αλλάζουμε τα επιχειρησιακά μας ε, σχέδια και τους στόχους μας. Δεύτερον, συζητούμε για δομικές αλλαγές με συγκεκριμένες ομάδες αφοσιωμένες στη στήριξη και στον συντονισμό τέτοιων προγραμμάτων. Γιατί για να πετύχουμε αυτό το 50% αυτό το φιλόδοξο στόχο χρειαζόμαστε κόσμο που να συντονίζει τα πράγματα και να είναι αφοσιωμένος ειδικά σε αυτό. Και τρίτον, όπως είπα, εκπονούμε αναθεώρηση για την επιλεξιμότητα βάση ε, της γραμμής των Παρισίων. Και γενικότερα την πολιτική μας θέλουμε να την ευθυγραμμίσουμε με τους περιβαλλοντικούς στόχους. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Φτάνουμε στο τέλος αυτής της συζήτησης που ήταν μια πλούσια συζήτηση, πολύ ενδιαφέρουσα. Και νομίζω εδώ ότι υπό το φως των όσων άκουσα σήμερα να επενθυμίσουμε και κάποια βασικά στοιχεία ε, που αφορούν την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η ΕΤΕΠ δημιουργήθηκε με τη συνθήκη της Ρώμης και στόχος της είναι να υλοποιεί τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων διασφαλίζεται από τις χώρες μέλη, που είναι και οι μέτοχοι της τράπεζας αυτής. Για τους υπόλοιπους, για μας εδώ στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, είναι πολύ σημαντικό να φροντίσουμε ώστε οι εγγυήσει και η πολιτική επενδύσεων ε, δικιά σας θα συνεχίσει να στηρίζει και να προωθεί τους στόχους της συνοχής. Δεύτερον, όσον αφορά το κλίμα. Ήδη κρατώ ότι το 2018 ήδη το 30% της πολιτικής σας ε, πηγαίνει ε, στο κλίμα. Και ο στόχος σας είναι ένας πολιτικός στόχος για παραπάνω. Κάτι το οποίο συζητιέται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που αποφασίζεται και στις χώρες μέλη. Και εφαρμόζει, υλοποιεί στη συνέχεια η ΕΤΕΠΑ. Συνεπώς, για την υλοποίηση αυτή είναι πολύ σημαντικό εμεί, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Επιτροπή Περιφερειακών Υποθέσεων που ασχολείται με τη συνοχή, να παρακολουθεί τα πράγματα. Γι' αυτό και σας ε, ζητώ να υπάρχει πράγματι παρακολούθηση και συνέχεια στο στόχο αυτό της συνοχής. Έχουμε συζητήσει εδώ στην Επιτροπή μας το σχέδιο Juncker. Πολλές ανησυχίες εκφράστηκαν όσον αφορά τους στόχους της συνοχής. Έγιναν συζητήσεις για το θέμα της γεωγραφικής κατανομής κλπ. κλπ. Όλες αυτές οι συζητήσεις ε, έγιναν και τακτοποιούνται μέσα στον ε, κανονισμό. Τώρα, μετά το σχέδιο Juncker είναι καλό να ξέρουμε ποια είναι η άποψη της ΕΤΕΠ. Και εδώ ίσως γραπτά θα μπορούσατε να μας απαντήσετε. Τώρα που πηγαίνουμε προς την Συμφωνία Πράσινης Ανάπτυξης να δούμε ποιος είναι ο δικός σας απολογισμός από το σχέδιο Juncker. Η συζήτηση αυτή λοιπόν πιστεύω ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και σίγουρα θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν ακριβείς και σαφής και πλήρης στις απαντήσεις σας. Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Ευχαριστούμε. Euh, Περνάμε στο επόμενο θέμα της σα διάταξης. Γνωρίζετε ότι στις 11-12 του 19 η διάσκεψη των Προέδρων ενέκρινε την εκπόνηση έκθεση πρωτοβουλίας της Επιτροπής ΕΚΟΝ με τίτλο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για το Συντονισμό των Οικονομικών Πολιτικών, ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2020. Μετά την έγκριση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τροποποίησε τον τίτλο της έκθεσης και αντικατέστησε την ετήσια επισκόπηση με μια στρατηγική επισκόπηση. Ε, στο καλό να πάτε και σας ευχαριστώ. Ε, κατά τη ε, συνεδρίαση της 19ης 12 του 19 οι συντονιστές τη Επιτροπής ΕΚΟΝ αποφάσισαν συνεπώς να ζητήσουν τροποποίηση του τίτλου ε, της έκθεσης πρωτοβουλίας και έχει ως εξή τώρα Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για το Συντονισμό των Οικονομικών Πολιτικών ετήσια στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξη για το 2020. Άρα, η πρόεδρος της Επιτροπής ΕΚΟΝ έστειλε επιστολή στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου όπου ζητούσε την αλλαγή του τίτλου σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για το θέμα αυτό και την έκθεση αυτή, η προθεσμία ε, κατάθεσης τροπολογιών έχει οριστεί στις 23 ε, Πρώτου, 6 ώρα το απόγευμα. Οι συντονιστές μας αποφάσισαν να αναθέσουν τη γνωμοδότηση στην κυρία Φραντσέσκα Ντονάτο, στην οποία δίνω μέσω στο λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω στα Ιταλικά. Και ευχαριστώ και σας Πρόεδρε και όλους τους συναδέλφους ε, που μου αναθέσατε αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης που για μένα είναι πραγματικά μεγάλη τιμή όσο και προνόμιο. Ζητώ συγγνώμη από όλους τους συναδέλφους ε, γιατί είναι πολύ σφιχτό το χρονοδιάγραμμα για τις ε, τροπολογίες. Δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Η Επιτροπή ΕΚΟΝ. Εμείς δεν είχαμε καμία δυνατότητα επιρροής και τροποποίησης των ε, προθεσμιών. Άρα θα μπω αμέσως στο θέμα, να σας πω ποια είναι τα βασικά σημεία της πρότασης γνωμοδότησής μου. Ε, ξεκινώ από μια διαπίστωση. Ε, έχει επιβράδυνση η ανάπτυξη που προβλέπεται για το 2020 σύμφωνα με όλους τους οικονομικούς αναλυτές και τους οικονομικούς δείκτες, όπως φαίνεται άλλωστε και από την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κρατώ λοιπόν ότι Μάλλον να το πω αλλιώ, θέλησα να εστιάσω στην ανάγκη παρέμβασης ακριβώς για να αναζωογονηθεί ε, η οικονομία η οποία βρίσκεται σε αποτελμάτωση. Πώς θα εκκινήσει στη την ανάπτυξη, τη μεγέθυνση της οικονομίας από τις πιο καθυστερημένες οικονομικά περιφέρειες. Ποιες είναι αυτές οι περιφέρειες όπου ε, υπάρχει, που υπάρχει μεγαλύτερη ανεργία και ε, η μεγαλύτερη ανάγκη επενδύσεων κυρίως ε, δημοσίων επενδύσεων, οι οποίες χρειάζονται οπωσδήποτε για να ε, δημιουργηθεί μια ανάπτυξη σε αυτές τις περιφέρειες που εμφανίζουν σημαντική καθυστέρηση σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ε, την κοινωνική ένταξη, για την επιχειρηματικότητα, ιδιαίτερα των νέων. Ένα άλλο σημείο πολύ σημαντικό στο οποίο επικεντρώνω τη γνωμοδότησή μου είναι ότι η πολιτική συνοχή είναι το βασικό εργαλείο και το τονίζω αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να φτάσουμε σε αυτούς τους στόχους της οικονομικής ανάπτυξης. Είναι μια ανάπτυξη ισορροπημένη ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Προς το σκοπό αυτό ε, θυμίζω για άλλη μια φορά πόσο μεγάλη σημασία έχει να εξασφαλίσουμε ε, τους απαραίτητους πόρους στον προεπολογισμό, στο επόμενο PDP, το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, στο κεφάλαιο που έχει να κάνει ε, με το Ταμείο Συνοχής. Θέλησα επίσης να αναφέρω πόσο σημαντικό είναι να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο ρόλο της οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την Ευρωζώνη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ιδιαίτερα στην Ευρωζώνη. Για, ε, για μένα θα πρέπει να φροντίσει και να προσέξει να μην ε, κινδυνεύσουν οι προκυκλικές πολιτικές. Τι εννοώ, όταν βρίσκεται σε αποτελμάτωση και ε, επιβράδυνση η οικονομία. Δεν θα πρέπει να ακολουθεί ε, αυτή την εξέλιξη η διακυβέρνηση, αλλά να την αντιστρέφει. Θυρούν πάρα πολύ αυστηρά τα κριτήρια ε, και τις υποχρεώσεις τις δημοσιονομικές, αλλά αυτό που χρειάζεται είναι δημόσιες επενδύσεις και διαρθρωτικές ε, μεταρρυθμίσεις. Ε, δεν διαφωνώ ε, ότι αυτά είναι σωστά, αλλά χρειάζονται δημόσιες επενδύσεις και επενδύσεις που να πιάνουν τόπο και να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των περιφερειών. Για να έχουμε μεγένθηση της οικονομίας, αύξηση του ΟΕΠ και τελικά μείωση των ανισοτήτων. Πρέπει λοιπόν να υποστηριχθεί η δημόσια επένδυση, ακόμα και εκεί που είναι πολύ αυστηροί οι δημοσιονομικοί κανόνες. Η οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να γίνεται πολύ καλύτερα ε, και να αντιμετωπίζει τις ασυμμετρίες που υπάρχουν στην Ευρωζώνη. Και όχι μόνο. αλλά και στους προπολογισμού και στη ε, ισοζύγια εμπορικών συναλλαγών. Οι κάποιες ε, χώρες έχουν υπερβολικά ε, πλεονάσματα στις εμπορικές τους συναλλαγές, τα οποία θα πρέπει να μειωθούν. Και αν χρειαστεί να προβλέπουμε και ειδικού μηχανισμούς που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωμη Τάξη και να τους κινητοποιούμε. Υπάρχουν κάποιες χώρες που είναι ήδη ελληματικοί οι προϋπολογισμοί τους και δεν μπορούν να αντιμετωπίζουν από μόνες τους δυσκολίες. Μια χώρα που δυσκολεύεται και έχει πολύ λίγους πόρους δεν μπορεί ε, να επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο. Δεν είναι σωστό αυτό ούτε οικονομικά ούτε επιστημονικά. Στη συνέχεια, ε, τι γίνεται με τη βιωσιμότητα της ε, οικονομικής ανάπτυξης. Μιλούμε συχνά για βιωσιμότητα από τη σκοπιά της οικονομίας ή του περιβάλλοντος, του κλίματος και ξεχνάμε την κοινωνική βιωσιμότητα που είναι πάρα πολύ σημαντική και αυτή. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με την αναδιανομή του πλούτου, του, των πόρων. Θα πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί και να αυξηθεί και η παραγωγικότητα όπως είδαμε ε, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετιών, όπου είχαμε αύξηση της παραγωγικότητας χωρίς αύξηση των μισθών σε πραγματικούς όρους, αυτό που ακολούθησε ήταν οικονομική κρίση. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε θέσεις εργασίας ε, σταθερές, ποιοτικές, οπωσδήποτε να στηρίζουμε την επαγγελματική κατάρτιση, την έρευνα, την παιδεία να προσπαθούμε να έχουμε και κάποιες ε, κοινωνικές ε, αντισταθμίσεις όπου αυτό χρειάζεται. Αυτά είναι τα βασικά σημεία του σχεδίου γνωμοδότησής μου. Θα πρέπει να κάνω και εγώ κάποιες τροπολογίες. Να σας πω ποιες είναι οι προθεσμίες Υπάρχουν κάποιες τροπολογίες που θέλω να κάνω, ε, όπου θα αναφέρομαι σε ένα πρόβλημα που μας έχει ήδη απασχολήσει. Ε, το σχέδιο επενδύσεων για τη βιώσιμη Ευρώπη είναι πολύ σημαντικό και θα καταλάβει και σημαντικό τμήμα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Αν δεν υπάρχει όμως ο κατάλληλος οικονομικός ιστός ε, που να απορροφά τις επενδύσεις αυτές, δεν θα μπορέσουμε να τις υλοποιήσουμε. Ούτε μόχλευση θα δούμε, ούτε τίποτα. ενώ τα διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, είτε πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, είτε για την ΕΚΤ, ε, αυτά τα όργανα ενθαρρύνουν ε, την ε, ανάπτυξη αυτή, αλλά θα πρέπει να ανταποκρίνονται και οι περιφέρειες για να υπάρχει ένα καλό επενδυτικό κλίμα και να μπορούν οι επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται. Χρειάζονται έργα υποδομών που δεν υπάρχουν, διάφορα άλλα μέσα και εκεί πρέπει να παρεμβαίνει η πολιτική συνοχής και οι δημόσιες επενδύσεις όπως είπαμε. γίνονται διάφορες αναλύσεις και από την ίδια την ΕΤΕΠ για ε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Ε, περίπου 500 δισεκατομμύρια έχουν κινητοποιήσει, αλλά τελικά 65 δισεκατομμύρια είναι οι, οι επενδύσεις που έχουν πραγματικά υπογραφεί. Και ο πρώην πρόεδρος κατά είναι, να απάντησε, ε, ότι ε, αυτά είναι ακόμα υποσχέσεις που δεν έχουν υλοποιηθεί. Και είναι μακράς πνοής αυτά τα έργα, μακροχρόνια. Γιατί η δημιουργία αυτού του έφορου εδάφους που χρειάζεται Και τέλος, ιδιαίτερη ε, προσοχή πρέπει να δοθεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στο επιχειρηματικό πνεύμα, ιδιαίτερα στις χώρες της Μεσογείου, που δυσκολεύονται να αξιοποιήσουν αυτές τις δυνατότητες, ε, γιατί είναι και υπερβολική η γραφειοκρατία. Και τελικά οι μικρομεσαίε επιχειρήσεις χρεοκοπούν μέχρι να βρουν το δίκιο τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το τμήμα της ευρωπαϊκής οικονομίας και δεν θα πρέπει να το αφήσουμε να χρεοκοπήσει γιατί αυτό θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο αυτή την επιβράδυνση και αποτελμάτωση της ε, οικονομικής ανάπτυξης. Για να κλείσω, απευθύνω μία πρόσκληση ε, ε, προς την Επιτροπή ΕΚΟΝ και στη συνέχεια προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε να ε, γίνουν πιο αποτελεσματικοί οι στόχοι της Ένωσης για την εδαφική συνοχή, τη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα και την κοινωνική, ομοιογενή ανταγωνιστικότητα και αναδιανομή του πλούτου. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση που κάνατε. Θα αφήσω το λόγο τώρα ε, στους σκιώδες. Καταρχήν ο Τόμας από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, Έχει περάσει η ώρα και το θέμα το οποίο συζητάμε είναι εξαιρετικά σημαντικό. Για το λόγο λοιπόν αυτό θα προσπαθήσω να περικόψω κάπως αυτά τα οποία είχα σημειώσει να σας πω. Καταρχήν αντιμετωπίζω πολύ θετικά την πρόταση γνωμοδότησης κυρίας Ντονάτο και να σας πω πως συμπεριλαμβάνει κάποια στοιχεία εξαιρετικά ε, πολύτιμα και νομίζω αποτελεί και τη σωστή βάση για να συζητήσουμε το θέμα αυτό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εδώ στο εσωτερικό της Επιτροπής μας. Δεύτερον, έχω διάφορα σχόλια τα οποία θέλω να κάνω. Ε, η συγγήτρια έχει βάλει πολύ θετικά στοιχεία μέσα και εμείς σε αυτά δεν έχουμε αντίρρηση. Αλλά κάποια από τα επιχειρήματα που αναφέρονται δεν θα έπρεπε να εμφανίζονται σε γνωμοδότηση της Επιτροπής ε, Ρέτζι, γιατί δεν είναι της δικής μας αρμοδιότητας. Είναι θέματα τα οποία, για τα οποία είναι αρμόδια άλλες επιτροπές, οπότε εμείς θα έπρεπε να εστιάσουμε σε αυτά τα οποία είναι πιο πολύ μέσα στο δικό μας χώρο. Για παράδειγμα, τα εμπορικά ζητήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά, δεν έχουν όμως χώρο εδώ. Δεν μπορούν να αποτελούν προτεραιότητα σε σχέδιο γνωμοδότηση της δικής μας επιτροπής. Όντως, Όντως, εδώ έχουμε το τεράστιο εργατικό δυναμικό της Ευρώπης, το οποίο θα πρέπει να προστατεύσουμε ε, μισθούς, ε, εργασίας. Δεν διαφωνώ, αλλά γιατί αυτό θα πρέπει να είναι κομμάτι γνωμοδότησης της δική μας Επιτροπής. Επίσης, παρόλο που συμφωνώ απολύτως και συμφωνούμε απολύτως με κάποια άλλα σημεία, ε, ίσως καλό θα ήταν κάποια επιχειρήματα να τα εντάξουμε αλλού το μόνο που έχω να σας πω είναι ίσως καταθέσουμε σχετικές τροπολογίες γιατί η ανεργία ναι, είναι ένα τεράστιο θέμα. Είναι πολύ ουσιαστικό. Θα πρέπει να μιλάμε για κοινωνική ένταξη, για ανεργία, για περιφερειακή πολιτική και πόσο η περιφερειακή πολιτική σχετίζεται και τι ρόλο καλείται να παίξει στη δημιουργία απασχόλησης και θέσεων εργασίας. Επίσης, το θέμα της μακροχρόνιας ανεργίας θα πρέπει να υπογραμμιστεί όπως επίσης και η ανεργία των νέων. Βεβαίως, είμαι μεγάλος και πια έχω αρχίσει να γίνομαι και απεσιόδοξος. Γιατί συνέχεια ζητάμε να μειωθεί το διοικητικό άχθος. Δεν πιστεύω πια ότι γίνεται αλλά πιστεύω ότι και η περιφερειακή πολιτική θα πρέπει να το επιδιώξει. Δηλαδή το διοικητικό βάρος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλό θα ήταν να μειωθεί. Δεν φτάνει να μιλάμε μόνο για το πόσο σημαντικέ είναι οι μικρομεσαίε επιχειρήσει στη δημιουργία θέσεων απασχόληση. Θα πρέπει να μειώσουμε και την ε, γραφειοκρατία, η οποία κάνει τη ζωή του δύσκολη. Και ένα σημείο αφετηρίας για το ΕΛΚ είναι οι πολιτικές ε, επενδύσεων ε, στην Ευρώπη να είναι πετυχημένες. Και εδώ συμπεριλαμβάνουμε και την περιφερειακή πολιτική. Αν βλέπουμε δηλαδή ότι λαμβάνουμε μηνύματα ε, πως επιβραδύνεται η οικονομία, η οικονομική ανάπτυξη, τότε θα πρέπει με τον προϋπολογισμό που έχουμε για την ε, ε, περιφερειακή πολιτική να βοηθήσουμε όσο μπορούμε έτσι ώστε να διατηρήσουμε το ρόλο μας που είναι αυτός της, του κινήτρου ε, που θα δώσει μια όθηση στην ευρωπαϊκή οικονομία. Μην ξεχνιόμαστε. Έχουμε το Green Deal και αυτό θα έχει πολλές επιπτώσεις στην οικονομική μας πολιτική. Αλλά μην νομίζετε πως κάθε φορά που λέμε Green Deal ή Πράσινο Σύμφωνο θα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ως ε, ένα μάντρα το οποίο θα λύσει ε, μια ευχή που θα λύσει όλα τα προβλήματα της Ευρώπης. Την ψηφιακή μεταρρύθμιση, την τεχνολογική προσαρμογή, την εφαρμογή ε, γενικότερα ε, των τεχνολογιών του 21ου αιώνα σε κοινωνικό επίπεδο. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία θα εμφανιστούν στις τροπολογίες που θα καταθέσει το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεισφορά αυτή. Σοσιαλιστές δεν βλέπω το σκιώδη ηγητή. Οπότε ο Έρικ Μπέρκβιστ από την ομάδα Renew. I will be... I will... Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Διάβασα την γνωμοδότηση της ε, ε συναδέλφου. Ευχαριστώ κύριε Αντωνάτο. Θα κάνουμε κάποιες τροπολογίες ε, για τις ε, πράσινες προτεραιότητες και τις κοινωνικές αλλαγές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε την πράσινη συμφωνία που θα φέρει αλλαγές που θα επηρεάσουν όλη την Ευρώπη. Όπως είπε και ο κύριος Ντόιτς, παντού υγεία, κοινωνικά, περιβαλλοντικά, οικονομικά, θέματα παιδείας. Όλες αυτές τις αλλαγές θα πρέπει να τις λάβουμε υπόψη και να τονίσουμε πόσο σημαντικό είναι να έχουμε καλές πολιτικές και μετρήσιμα στοιχεία. Είναι καμπή, θα μπορούσαμε να πούμε, για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες σήμερα και πρέπει όλα να τα λαμβάνουμε υπόψη. Σας ευχαριστώ. Merci beaucoup, Vlad ευχαριστώ πολύ κύριε Μπότος. Από την ΚΟΕ η Μαρτίνα Μίχιλς κάθεται εκεί αλλά δεν θέλει να μιλήσει. Ωραία. Ε, ο συνάδελφος Μπούντα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ομολογώ ότι έχει περάσει καιρός από τότε που έχω να δω μια τόσο ολοκληρωμένη γνωμοδότηση. Η συνάδελφος έχει εντοπίσει σωστά πάρα πολλά σημεία. Καμιά φορά, όπως είπε ο κύριος ε, Ντόιτς, ε, ξεπερνάμε τις αρμοδιότητές μας, αλλά δεν μπορούμε να αγνοούμε αυτά τα πράγματα και θα πρέπει να τα γράφουμε στις γνωμοδοτήσεις γιατί είναι αλληλένδετα. Ε, εμείς συζητούμε για την πολιτική συνοχή. Αυτή επηρεάζει καθημερινά τη ζωή μας. συζητούμε για την απλούστευση, ότι είναι κάτι ε, το οποίο μας ενδιαφέρει πολύ. Από τότε που έχω έρθει στο Κοινοβούλιο, πάνω από έξι χρόνια πριν, ακούω για απλούστευση. Ε, ότι εάν είναι πιο απλή στη διαχείριση, η διαχείριση μπορούν τα κονδύλια να αξιοποιούνται καλύτερα. Ε, είναι πολύ περίπλοκοι οι κανόνες, γι' αυτό οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δυσκολεύονται να χρηματοδοτηθούν. Ακούστηκε και το θέμα της ανεργίας. Είναι γεγονός ότι υπάρχει ανεργία παντού. Υπάρχουν όμως και κάποιες περιφέρειες και αυτό θα πρέπει να το γνωρίζουμε. Ιδιαίτερα στην Ανατολική Ευρώπη, όπου δεν έχουμε αρκετά εργατικά χέρια για να εφαρμόζουμε τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Τι μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχουν χώρες όπως η Ρουμανία και η Βουλγαρία που μπορεί να έχουν πολλούς οικονομικούς πόρους στη διάθεσή τους από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Δεν έχουν αρκετούς εργαζόμενους για να τα αξιοποιήσουν. Και άμα δεν τα αξιοποιήσεις δεν μπορείς να αναπτύξεις ε, τις τοπικές κοινωνίες και οι τοπικές κοινωνίες αισθάνονται καταλελειμμένες και ο κόσμος μεταναστεύει στην εσωτερική εξωτερική μετανάστευση. Θα πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη μας, ότι ο κόσμος φεύγει και πώς θα το κρατήσουμε στον τόπο του τον εργαζόμενο ε, για να βρούμε κάποιους μηχανισμούς και τρόπους ακόμα και να ξαναγυρίσουν όσοι έχουν φύγει και να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της τοπικής τους κοινωνίας. Αλλιώς θα έχουμε περιφέρειες ακατοίκητες τελείως και στο μέλλον θα είναι πολύ δύσκολο να φέρουμε νέο πληθυσμό. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. Ευχαριστούμε πολύ. Καλώς. Ευχαριστώ λοιπόν τις πολιτικές ομάδες που συμμετείχαν στη συζήτηση αυτή και παρουσίασαν τις θέσεις τους σε σχέση με την εισηγήτρια την κυρία Ντονάτο, προθεσμία για υποβολή τροπολογιών είναι 23 23η Ιανουαρίου στις 6 το απόγευμα. Ολοκληρώνεται λοιπόν το σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη και περνάμε στο επόμενο σημείο που είναι ένα σημαντικό σημείο και το οποίο αφορά την έκθεση που πρέπει εμείς να εκπονήσουμε εδώ στην Επιτροπή μας όσον αφορά ε, τις ε, συζητήσεις και τους τριμερείς διαλόγους που λαμβάνουν χώρα σε σχέση με τον κανονισμό για την συνοχή. Ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μας υποχρεώνει να ε, παρουσιάσουμε έκθεση στην Επιτροπή μας. Και αυτό ακριβώς κάνουμε τώρα. Και υπενθυμίζω επίσης ότι η Φιλανδική Προεδρία από τη δικιά της την πλευρά παρουσιάζει στο κοινό την κατάσταση των διαπραγματεύσεων όπως αυτές έχουν προχωρήσει μέχρι σήμερα. Υπενθυμίζω λοιπόν ότι στο δεύτερο εξάμενο του 2019 οι τριμερείς διάλογοι για τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων ξανάρχισαν και έγιναν τρεις την προηγούμενη θητεία υπό Ρουμανικής Προεδρίας και είχαμε και τρεις νέους υπό φιλανδική προεδρία. Ο τέταρτος τριμερής διάλογος έλαβε χώρα στις 3 Οκτωβρίου, ο πέμπτος στις 12 Νοεμβρίου, ο έκτος στις 27 Νοεμβρίου και έβδομος στις 10 Δεκεμβρίου. Εκ παραλίλου με τους διαλόγους αυτούς έγιναν και διάφορες τεχνικές συναντήσεις και υπήρξαν και άτυπες επαφές. φτάσαμε στην 10η Δεκεμβρίου και προσέξτε σε μια κοινή προσωρινή κατανόηση με το Συμβούλιο όσον αφορά τα τμήματα 1, 2 και 5. Η Κορεπέρα από τη δικιά της την πλευρά επιβεβαίωσε ότι αυτή η κοινή προσωρινή κατανόηση της 18 Δεκεμβρίου του 2019 δημοσιεύθηκε από τη Φιλανδική Προεδρία λίγες μέρες μετά τη συζήτηση στην Κορεπέρ. Υπενθυμίζω ότι τα όσα συμφωνήθηκαν παραμένουν προσωρινά και τίποτα δεν συμφωνείται εφόσον δεν έχουν συμφωνηθεί όλα βάσει της γνωστής αυτής σε όλους αρχής. Ο κανονισμός περί κοινών διατάξεων και ο πιο δύσκολος που διαπραγματευόμαστε εμείς είναι 112 άρθρα, 180 σελίδες για να συντονίσουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής, το Interreg, το Ταμείο για την Μετανάστευση, για την Εσωτερική Ασφάλεια κλπ. κλπ. Όπως επίσης και ένα εργαλείο για την διαχείριση των συνόρων. Πρόκειται λοιπόν για έναν πολύ βασικό κανονισμό για περισσότερο από το 1 τρίτο του μελλοντικού προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είχα την ευθύνη να προεδρεύσω αυτών των τριμερών διαλόγων και θέλω να συγχωρώ εδώ τον κύριο Νόβακοφ και Σκλέλ, τους συνεισηγητές, για το έργο τους. Τους ευχαριστώ επίσης, όπως και τις διάφορες αρχές, για την συμμετοχή τους. Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες τώρα για όλα τα επεισόδια τα οποία έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Πάντως οι συνεισηγητές κατάφεραν ανα πάσα στιγμή να κάνουν θετικές προτάσεις και τολμηρές θα έλεγα, οι οποίες απέτρεψαν να καταλήξουμε στο συμπέρασμα που θα σας παρουσιάσουν. Συνεπώς, τους δίνω και το λόγο για λίγα λεπτά και θα συζητήσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες τι πέτυχε τελικά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πιο συγκεκριμένα για το ΦΕΝΤΕΡ το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ξεκίνησε σε αυτή τη θητεία ο διάλογος και στις 12 Δεκεμβρίου έγινε αυτός. Με συζητήσεις για το ΕΤΠΑ που ήταν πολύ πυκνές μέχρι τώρα, δεδομένου ότι το άρθρο βρίσκεται στο διαπραγματευτικό κουτί του Συμβουλίου και έχει αντίκτυπο σε διάφορα άρθρα του κανονισμού και το Συμβούλιο δεν θέλει να προχωρήσει πολύ. Πάντως, έστω η περιθεριακή ε, πρόοδος που έγινε είναι πραγματικότητα και εδώ χαιρετίζω το έργο του Αντρέα Κοτσολίνο, του εισηγητή μας, που σε λίγο θα μας παρουσιάσει το κομμάτι που αφορά το ΕΤΠΑ. Και όσον αφορά το Ιντερεκ, ο Πασκάλα Ριμό, ελπίζω ότι θα επανέλθει για να μας το παρουσιάσει. Είχαμε τρεις τριμερείς διαλόγους, Νοεμβρίου και 10 Δεκεμβρίου. Εδώ το έργο ήταν πολύ σημαντικό για το μισό περίπου κανονισμό, εξού και ευχαριστώ πολύ τον Πασκάλα Ρημό για, το... για την προσπάθειά του και θα μας τα εξηγήσει σε λίγο. Οπότε ζητάω από τους συγητές να παρουσιάσουν την πρόοδο που πετύχαμε, όπως επίσης και τα εκκρεμούντα θέματα στις ε, διοργανικές διαπραγματεύσεις για τους νομοθετικούς φακέλους που εξετάζουμε. Παρακαλώ ε, τους συζητητές να μην μας παρουσιάσουν σήμερα το αντικείμενο των ε, συζητήσεων που θα ακολουθήσουν, γιατί αυτό θα συζητηθεί με τους συντονιστές σε λίγο. Οπότε, Αντρέιν Νόβακοφ πρώτα. Και μετά, ε, κυρία Κρέλ, Κωνσταντ Κρέλ για τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για τα ευγενικά σας λόγια και για την εκτίμηση που δείξατε για όλη τη σκληρή δουλειά που κάναμε για αυτές τις ε, κοινέ διατάξεις και η Κωνσταντσα και εγώ, γιατί κάναμε πολλές προσπάθειες από κοινού, κράτησαν γύρω στα δύο χρόνια και νομίζω ότι έχουμε καλύψει το ίμιση του κανονισμού ε, στα πλαίσια της Φιλανδικής Προεδρίας. Ήταν πολύ δύσκολη η προσπάθεια αυτή, κυρίως λόγω της ε, μεταλασόμενης άποψης του Συμβουλίου, αλλά όχι μόνο. Ξέρω πως ε, στις τρέχουσες συνθήκες και για τη θέση του Συμβουλίου για τις πολιετής δημοσιονομικές προοπτικές, χρειάζεται και να αλλάξουμε προσέγγιση για να στείλουμε ένα μήνυμα και νομίζω ότι μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό χωρίς να ακυρώσουμε απολύτως την διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Δηλαδή, ε, συναντήσεις σε επίπεδο τεχνικών ε, θεμάτων για να κλείσουν τεχνικά ζητήματα ε, τα οποία το επόμενο διάστημα θα βοηθήσουν πάρα πολύ τον τριμερή διάλογο. Διαφορετικά, ό,τι έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα, Ό,τι έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα λοιπόν να το αφήσουμε στην άκρη και να ξεκινήσουμε ε, πάλι από την αρχή δεν είναι η σωστή τακτική και δεν θα ήθελα εγώ να συμβεί κάτι τέτοιο. Ξέρω πως δεν μπορούμε να προχωρήσουμε με την ίδια ταχύτητα, αλλά πιστεύω πως μπορούμε να κάνουμε αργή και σταδιακή πρόοδο, περιμένοντας να δούμε ποια θα είναι η θέση του Συμβουλίου για τις Πολιτικές ε, προοπτικές και κυρίως υπογραμμίζοντας πως εμείς δεν θα εγκαταλείψουμε τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Euh, Ευχαριστώ. Σας υπενθυμίζω. Το σημείο αυτό είναι στην ημερήσια διάταξη με τυπικό τρόπο πάντα για να ενημερώσουμε ε, την Επιτροπή για το πώς τρέχουν οι διαπραγματεύσεις. Άρα λοιπόν μπορούμε να μπούμε και λίγο σε λεπτομέρειες για τα όσα συνέβησαν και το τι οδήγησαν σε αυτή την ε, ε, προσωρινή κοινή συμφωνία για τα θέματα από το 1 μέχρι το 5. Εμείς εδώ δεν είμαστε και κλεισμένων των θυρών. Έχουμε εδώ πέρα και προσκεκλημένους, έχουμε και την Κομισιόν και το Συμβούλιο και κάποιες άλλες οργανώσεις, όπως επίσης και τον τύπο, οι οποίοι μας ακούν. Οπότε θα αφήσουμε ε, τα θέματα τα πιο στρατηγικά στην άκρη για το πώς πρέπει να προχωρήσουμε από εδώ και στο εξής. Θα δώσω τώρα το λόγο στην ε, Κωνσταντσα για να μας κάνει και αυτή τη δική της ενημέρωση. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. κάτι αντιχούσε, αλλά τώρα νομίζω είναι καλύτερα. Ε, θα πρέπει λίγο να το συζητήσουμε. Πρώτον, τι αποφασίσαμε και ποιος ήταν ο στόχος. Δεν ξέρω γιατί έχει τέτοια αντίχηση εδώ πέρα. Τι κάνω. Keine Ahnung. Ναι. Ξέρω τώρα έφτιαξε. Ναι, τώρα σε ακούμε πολύ καλά. Εγώ ακούω μια εχώ εδώ πέρα. Τι να κάνω. Ε, ε, στη φιλανδική Προεδρία θέλαμε να κλείσουμε τις ενότητες 1, 2 και 5. Αυτά τα μπλοκ που είναι απαραίτητα έτσι ώστε να μπορέσουν οι, οι περιφέρειες να αρχίσουν τον προγραμματισμό των ε, επιχειρησιακών σχεδίων, τα ΕΣΠΑ. Ε, δεν ήταν καθόλου εύκολο αυτό, γιατί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στις διαπραγματεύσεις ήταν ότι ορισμένα κράτη-μέλη αγωνίστηκαν να μην υπάρχουν στο μέλλον καθόλου εταιρικέ συμφωνίες. Περίεργο λίγο, γιατί σε αυτή την προγραμματική περίοδο αυτό θεωρήθηκε μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή, να έχουν μια στρατηγική εικόνα τα κράτη και ήταν υποχρεωμένα να το αναπτύξουν αυτό και αυτό έχει νόημα πραγματικά αν θέλεις να έχεις μια πολιτική ε, συνοχής στοχευμένη και με στοχό προσήλωση. Για μας το Κοινοβούλιο αυτό ανέκαθεν ήταν πάρα πολύ σημαντικό και ουσιώδους σημασίες και με την αρχή της εταιρικής σχέσης. Δηλαδή, ε, να μην έχουμε μόνο υπαλλήλου ε, από τα Υπουργεία που να συνεννοούνται, αλλά είναι και οι κοινωνικοί εταίροι, παραγωγικές τάξεις, η τοπική πολιτική, ε, περιβαλλοντικές οργανώσεις, άλλες μεγάλες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε μια περιφέρεια να συμμετέχουν και στη συζήτηση για το πού θέλει να πάει κάθε περιφέρεια. Εμείς καταφέραμε να βρούμε ένα συμβιβασμό τελικά που αλλάζει λίγο τη στρατηγική προσέγγιση. Αλλά για κράτη-μέλη που έχουν ένα μόνο ταμείο ή που παίρνουν λίγα χρήματα, ε, απλουστεύει πάρα πολύ τη ζωή τους. Ε, και μπορούν να το γράψουν αυτό και σε ένα χαρτί και να προχωρήσουν με τα ΕΣΠΑ και να τα υποβάλουν από κοινού. Προς μεγάλη μας χαρά επίσης καταφέραμε να επιβάλλουμε σημαντικά θέματα στις λεγόμενες οριζόντιες αρχές που τις έχουμε κατοχυρώσει. Μπορεί να θυμάστε ότι είχαμε συζητήσει πάρα πολύ εδώ στην Επιτροπή μας. Ήταν και πάρα πολλές οι για κάποιες οριζόντιες ε, σκέψεις στον συνολικό κανονισμό, όπου εμείς ως συνεισηγητές αποφασίσαμε να υποβάλουμε στην Επιτροπή μας μία δέσμη ενιαία. Αυτό δεν άρεσε στα κράτη-μέλη ούτε στην Προεδρία. Γιατί θεώρησαν ότι ήταν άχρηστα και περιτά αυτά που προτείναμε. Εν πάση περιπτώσει το περάσαμε, καταφέραμε να το επιβάλλουμε. Για την κλιματική αλλαγή και κάποια άλλα σημεία καταφέραμε να τα περάσουμε, παρά το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη τα είχαν κοινώς στη Ε, για την πρώτη ενότητα, συμφωνήσαμε για τον κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος καθίσταται πλέον απαραίτητος και πρέπει να προσαρμοστεί και στο νέο κανονισμό, αλλά τελικά βρέθηκε ένας δρόμος ανάμεσα στις τρεις νομικές υπηρεσίες των θεσμικών οργάνων, έτσι ώστε να είναι πολύ απλή η προσέγγιση και είναι μια απλή προσαρμογή, ας πούμε, στις αλλαγές που προκύπτουν με το νέο κανονισμό δεν έχουμε εκπώνηση από την αρχή με νομοθετική διαδικασία κλπ. Επίσης είναι πολύ σημαντικό αυτό για τις περιφέρειες. Τι άλλο. Στα ζητήματα της τεχνικής υποστήριξης και βοήθειας από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, περάσαμε τη δική μας θέση και ανταυτού δεχτήκαμε βέβαια τα κράτη-μέλη να κάνουν κάποιες αλλαγές ενδεχομένω. Αυτό που είχε για μας σημασία είναι να διευκρινιστεί το ζήτημα του ελέγχου. Δηλαδή, τα κράτη-μέλη που συνεργάζονται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να έχουν πιο απλές διαδικασίες σε σύγκριση με κάποια άλλα κράτη-μέλη που δεν συμμετέχουν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Καταφέραμε να το περάσουμε αυτό σε ένα συμβιβασμό και να το επιβάλλουμε. Και στις δημόσιες προμήθειες επίσης πετύχαμε μια σειρά από συμβιβασμούς αμοιβαίω υποφελή. Και αυτό ήταν σημαντικό και για τα τρία όργανα, όχι μόνο για τα δύο, και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάπου βρήκαμε ένα τρόπο και ένα δρόμο συνεννόησης και καταλήξαμε και σε αυτό. Προσωπικά πιστεύω ότι το αποτέλεσμα είναι συμβιβασμός, όπου έμειναν δυσαριστημένες όλες οι ε, πλευρές, άρα πρέπει να προσθέσω ότι είναι μάλλον καλό ο συμβιβασμός όταν δεν πολύ αρέσει σε κανέναν. Να το πω αλλιώ, το Κοινοβούλιο σε κάποιες περιπτώσεις θα μπορούσε να έχει επιβάλει περισσότερα. Η ηλεκτρονική συνοχή γιατί παραμένει εξαίρεση για ορισμένα κράτη-μέλη. Αυτό πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Αλλά αν αυτό ε, ε, βοήθησε να βρεθεί συμβιβασμό, άξιζε τον κόπο να το απεμπολίσουμε για να επιτύχουμε αυτό το συμβιβασμό. Και τελικά, εσπίσμα όλων των ε, προσδοκιών στις 10 Δεκεμβρίου καταφέραμε να συμφωνήσουμε σε ένα συμβιβασμό. Είναι σημαντικό μήνυμα και σημαντικό σημάδι και η τώρα Προεδρία, ποια είναι η Κροατική, θα πρέπει να βρει ένα δρόμο να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Θα εξαρτηθούν πολλά από τον τρόπο με τον οποίο θα φερθεί το Συμβούλιο για το PDP, οποίο και αν κάνει τις διαπραγματεύσεις. Αυτό θα φανεί τις επόμενες εβδομάδες και θα τα ξανασυζητήσουμε. Για τις περιφέρειες πάντω έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα. Υπάρχει τώρα ένας βασικός σκελετός που καταλαβαίνουμε τι πάνω κάτω σημαίνει και θα πρέπει να γεμίσει τώρα το υπόλοιπο οικοδόμημα. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Συμμερίζομαι απόλυτα την απόψή σου. Πιστεύω ότι η κοινή προσωρινή κατανόηση, ο συνολικός συμβασμός, είναι ένας συμβιβασμός ο οποίος ελάχιστα απομακρύνεται στην πραγματικότητα από την εντολή που λάβαμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και όσον αφορά τα ουσιώδη, τις αρχές που καθορίσαμε στην αρχή, μας ικανοποιεί. Πάντα βέβαια μέσα σε ένα πνεύμα συμβιβασμού, έτσι. Τώρα, επί του παρόντος, το μπαλάκι είναι στην κρατική Προεδρία. Γιατί πρέπει επίσης να πούμε ότι το negotiating box, το διαπραγματευτικό κουτί, είναι κάτι που εμπόδισε την καλή πρόοδο του διαλόγου. Οπότε ελπίζουμε το πνεύμα της Προεδρίας του Συμβουλίου να εξελιχθεί, αλλιώς θα είναι πολύ πιο δύσκολο Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο τώρα στον συνάδελφο Κοτσολίνο για να μας μιλήσει για τις διαπραγματεύσεις όσον αφορά το ΕΤΠΑ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Όντως και το ΕΤΠΑ υποφέρει από αυτό το γενικό κλίμα. Στη Ρουμανική Προεδρία δεν συγκλήθηκε καν ο τριμερής ε, διάλογος, ούτε τεχνικές συναντήσεις. Επί Φιλανδικής Προεδρίας, ναι. 12 Δεκεμβρίου, στα τέλη της χρονιάς, ε, ξεκινήσαμε να δουλεύουμε πάνω στο άρθρο αυτό, το 1α, 2, ε, αδιέξοδο στο 3 ό,τι έχει να κάνει με το δημοσιονομικό πλαίσιο. Ε, προχωρήσαμε στο 2, αλλά τίποτα ουσιαστικό. Τώρα λοιπόν πρέπει να δούμε πώς θα συνεχίσουμε με την ε, Κροατική Προεδρία. Κάπως ξεκίνησαν τα πράγματα, 9 Ιανουαρίου. Περιμένουμε να υπάρξουν και πολλές δραστηριότητες κάθε εβδομάδα τεχνικές συναντήσεις. Χρειάζεται μια γενική πλαισίωση βέβαια. Ορισμοί αποφάσεις και ίσως να συγκληθεί και τριμήρης διάλογος για το άρθρο 3 που είναι σημαντικό, τη θεματική συγκέντρωση και για το σημείο 6 επίσης. Μετά την ψηφοφορία στην Ολομέλεια Το είπε και ο κύριος ε, Σασόλη ότι πρέπει να διευκρινιστούν περισσότερα τα πράγματα. Πήραμε και κάποιο σημείο μου από αυτόν. Είναι ζωτική σημασία πάντω για το ΕΤΠΑ. Τώρα περιμένουμε τις πολιτικές αποφάσεις. Και μετά θα δούμε πώς θα συνεχίσουμε με τεχνικές συναντήσεις, με σύγκληση νέων τριμερών διαλόγων υπό Προεδρίας. Αυτό είναι το έργο μας πάντως. Ευχαριστούμε πολύ, λέει Ευχαριστούμε, Αντρέα. Πράγματι, θα δούμε για το ΕΤΠΑ. Ποια θα είναι η τοποθέτηση της κρατικής Προεδρίας, κυρίως για τα ουσιώδη άρθρα. Εφόσον μέχρι τώρα ήταν εκτός τριμερούς διαλόγου. Τώρα, ο Πασκάλ Λαριμό δεν είναι εδώ για το Interreg. Εγώ θα σας πω ότι για το Interreg πετύχαμε σημαντική πρόοδο για πολλά άρθρα του κανονισμού. Πάντως για το Interreg το βασικό πρόβλημα είναι πρόβλημα χρηματοδότησης. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε να βρούμε συμφωνία. Υπάρχει διάθεση από το Συμβούλιο, αλλά εμείς έχουμε πρόβλημα με το οικονομικό σκέλος. Και συνολικά για τον κανονισμό μας είναι πράγματα που δεν μπορούν να βγούνε από την γενικότερη διαπραγμάτευση που γίνεται σήμερα με το Συμβούλιο για τις Κοινέ Διατάξεις. Εξού και υπάρχει ένα συνολικό πλαίσιο συζήτησης και διαβούλευσης μεταξύ των εισηγητών, συνεισηγητών και από την πλευρά των συνεισηγητών ε, της Επιτροπής Προϋπολογισμών, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε συντονισμένα. Γιατί μπορούμε να έχουμε τον καλύτερο δυνατό κανονισμό, αν όμως δεν έχουμε ε, τον αντίστοιχο προπολογισμό, δεν θα πετύχουμε τους στόχους μας. Όπως και να έχει το πράγμα πάντως, η Επιτροπή μας ήταν παρούσα για να ανταποκριθεί και στο αίτημα των περιφερειών και ποιο είναι αυτό? Ο κανονισμός κοινών διατάξεων πρέπει να επιτρέπει στις περιφέρειες να δημιουργήσουν το νέο πλαίσιο κάτω από τις καλύτερες δυνατόν συνθήκες χωρίς καθυστερήσεις. Οπότε, σας ευχαριστώ για τις διευκρινήσεις σας. Οπότε κλείνει η κύρια συνεδρίαση της Επιτροπής μας εδώ και σας υπενθυμίζω ότι θα συνεχίσουμε αύριο, όχι στις 9, αλλά στις 9 και 30. Και στη συνέχεια θα έχουμε τη συζήτηση με την Επίτροπο Φερέιρα στις 10. Σας ευχαριστώ πολύ. Όσοι δεν πρέπει να είναι εδώ για τη συνεδρίαση των συντονιστών, παρακαλώ να βγουν από την αίθουσα. Ισύχως όμως. Εμείς θα συνεδριάσουμε με τους συντονιστές σε 15 λεπτά. Και ευχαριστώ και τους διερμηνείς για τις εξαίρετες υπηρεσίες τους. Ευχαριστούμε πολύ. Σε 15 λεπτά θα συνεχίσουμε για τη συνεδρίες των συντονιστών. Ευχαριστώ.